Okay, um, <clears throat> Καλημέρα σε όλους και σε όλες. <clears throat> Ξέρω ότι έχουμε καθυστερήσει λιγάκι. Αλλά είχαμε ε, να συζητήσουμε για τη διαδικασία που θα ακολουθήσουμε σήμερα το πρωί. Η πρόθεσή μας ήταν στην αρχή να έχουμε μια συνάντηση με την κυρία Έλενα Σαλγάδο, την πρόεδρο του Euro <clears throat> του ΕΚΟΦΗΝ. Την είχαμε προσκαλέσει βάσει των, την είχαμε καλέσει βάσει των νέων εξουσιών που έχουμε με τη της Λισαβόνας. Δυστυχώς χρειάστηκε να αναβληθεί και πάλι η έλευσή της εδώ. Ως εκ τούτου, <clears throat> επειδή πολλά μέλη είχαν πει ότι θα χρειαζόμασταν χρόνο να κάνουμε μια συζήτηση για τα θέματα που έχουν να κάνουν με την οικονομική εποπτεία και με την παρακολούθηση των δράσεων που έχουν να κάνουν με τη διάσωση της Ελλάδος, είχαμε πει ότι θα χρησιμοποιήσουμε το χρόνο μας για να συζητήσουμε αυτά τα θέματα. Μπορώ να σας κάνω τώρα μια σύντομη σύνοψη της κατάστασης. Την προηγούμενη Κυριακή προχθές, οι Υπουργοί Οικονομικών ενέκριναν το μηχανισμό βοήθειας προς την Ελλάδα βάσει το των κανόνων που είχαν ήδη διατυπώσει το πρόγραμμά του Ένα κοινό πρόγραμμα τριετέ Ευρωπαϊκή Ένωση, διεθνέ Νομισματικό Ταμείο αποφασίστηκε, δίνει 110 δισεκατομμύρια ευρώ για να βοηθηθεί η Ελλάδα να μπορέσει να καλύψει τι ανάγκες χρηματοδότησής της για ένα τριετές χρονικό διάστημα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση συμβάλλει με 80 δισεκατομμύρια ευρώ, οι χώρες της ζώνης του ευρώ, εκ των οποίων μέχρι 30 θα δοθούν στο πρώτο χρόνο Τώρα, η εξάρτηση αυτής της χρηματοδότησης θα ενσωματωθεί σε απόφαση του Συμβουλίου βάσει των άρθρων 126 και 136 της Συνθήκης που θα πρέπει να εγκριθούν επίσημα από το Συμβούλιο Ακοφήν στις επερχόμενες μέρες. Ζητήσαμε καταρχήν από την κυρία Σαλγκάδο να έρθει ενώπιόν μας επί τη βάση των ε, συστάσεων πολιτικής που ενεκρίθησαν από το ΕΚΟΦΗΝ στις 16 Φεβρουαρίου του ενεστώτος έτους. Και βέβαια από τότε τα πράγματα έχουν εξελιχθεί σημαντικά. Είναι κάπως ε, <clears throat> ξεπερασμένη αυτή η δήλωση του ΕΚΟΦΗΝ του Φεβρουαρίου. Κάτι το για το οποίο εγώ λυπάμαι είναι ότι όταν έστειλα αυτή την πρόσκληση στην κυρία Σαλκάδο, αμέσως μετά από την έγκριση αυτής της σύστασης το Φεβρουάριο, και τώρα φυσικά είναι Μάης, δεν έχει καταστεί δυνατό ακόμα να έλθει ενώπιόν μας η κυρία Σαλγάδο. Και μου φαίνεται όχι ιδιαίτερα πρέπον το ότι οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβούλιου και ιδίω τη Επιτροπή μα είναι υποχρεωμένοι να πληροφορούνται από τα μέσα ενημέρωση και από το τύπο και όχι να έρχεται ενώπιον του το αρμόδιο το αρμόδιο μέλος της Ισπανικής Προεδρίας για να τους εξηγήσει περί τίνος πρόκειται. Είχαμε πει ότι θα μπορούσε να είναι και κλεισμένο των θυρών η συνάντησή μας με την κυρία Σαλγάδο και να υπάρχουν συμφωνίες για το τι μπορούμε να συζητήσουμε ή, ή όχι. Πάντως είπε η κυρία Σαλγάδο ότι δεν μπορεί να έρθει προς το παρόν και εμείς εξετάζουμε τη δυνατότητα να έρθει κατά τη διάρκεια της εβδομάδας του Στρασβούργου στις 17 ή στις 20 του μηνός. Συνεχίζοντας λοιπόν, <clears throat> ξέρουμε ότι τη Δευτέρα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αποφάσισε να δώσει μια ειδική μεταχείριση στα ε, ελληνικά ομόλογα υπομορφή εγγυήσεων και ο κύριος Φων Ρομπέι έχει ζητήσει από του αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων της περιοχής του ευρώ να παρακαθίσουν σε ένα δείπνο στις 7 Μαΐου, την Παρασκευή δηλαδή, για να λάβουν υπόψη, για να συζητήσουν μάλλον για τι κοινοβουλευτικέ διαδικασίες οι οποίε χρειάζεται να τεθούν σε κίνηση για να εγκριθεί η εκταμείευση των ποσών αυτών για την Ελλάδα. Επιπλέον, στο φω αυτή τη κρίση υπάρχει η πρόθεση να υπάρξει μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων σε σχέση με τα διδάγματα τα οποία πρέπει να αποκομίσουμε στην περιοχή του ευρώ, ιδίως ό,τι αφορά στην οικονομική διακυβέρνηση. Και από ό,τι κατανοώ, η πρώτη συνάντηση τη ειδική μονάδα που έχει θεσπιστεί από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο <clears throat> το Μάρτιο του ενεστώτος έτου για τα οικονομικά θέματα και τη διακυβέρνηση θα συναντηθεί αυτή η ομάδα για πρώτη φορά στις 21 Μαΐου. Η ομάδα αυτή θα αποτελείται κυρίως από υπουργού Οικονομικών και πρέπει να σα πω και πάλι ότι ο ρόλος του Κοινοβουλίου δεν έχει διαλευκανθεί. Έχουμε κάποιες πρόσθετες αρμοδιότητες και ευθύνες βάσει της νέας συνθήκης της Λισαβόνας και παρά τα αιτήματά μας προς το παρόν μας παραγνωρίζουν, για να μην το πω χειρότερα. Και όπως γνωρίζετε η Επιτροπή μας έχει ξεκινήσει κάποιες πρωτοβουλίες για ακροάσεις που έχουν εξετάσει κάποια από τα συναφή θέματα και νομίζω ότι φαίνεται ότι το έχουμε κάνει αυτό με έναν τρόπο ο οποίος ήταν απόλυτα υπεύθυνο. Είδαμε πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τον οικονομικό συντονισμό, την εποπτεία και τη διαχείριση των κρίσεων και να ενισχύσουμε την εποπτεία των χρηματαγορών, τη ρύθμιση, τη διαχείριση των κρίσεων και να βελτιώσουμε την αξιοπιστία των στατιστικών μας στοιχείων. και φυσικά μας απασχολεί και το γενικότερο έργο μας σε σχέση με την μελλοντική δομή που θα πρέπει να έχει υποπτία των τραπεζών και χρηματαγορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ως Νούπο θα ξεκινήσουμε και το έργο μας για την εφαρμογή των νέων ελεγκτικών εξουσιών της Eurostat. Αλλά πρέπει να διαδραματίσουμε και ένα σημαντικό ρόλο στη συζητήση για την οικονομική διακυβέρνηση και θα πρέπει να προσπαθήσουμε να έχουμε μια στεναρή θέση μέχρι το τέλος του χρόνου μεταξύ των μελών της Επιτροπής μας. Ελπίζω λοιπόν ότι και αυτή η ευκαιρία θα είναι πρόσφορη για να ξεκινήσουμε μια άτυπη ανταλλαγή απόψεων σε σχέση με τα διδάγματα τα οποία μπορούμε να αντλήσουμε από την κρίση και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. Αυτό λοιπόν το γενικό πλαίσιο και με μεγάλη χαρά μπορώ να δώσω τώρα το λόγο σε αυτούς οι οποίοι θέλουν να λάβουν το λόγο. Έχω στον κατάλογο μου τον Γκοζές, τον ε, Γκαρσία Μαργκάγιο. Ναι, βλέπω τώρα πολλά χέρια τα οποία σηκώνονται. Σβέν, η Περβάνς, ο κύριος Χουντής, Ποδηματά. Σίγουρα θα έχουμε καιρό να ακούσουμε όλες τις απόψεις. Ο Ζωάν Πολ πρώτα. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Πολύ σύντομα. Ήθελα να σας πω ότι συμφωνούμε απόλυτα με αυτά που είπατε και για το ότι θλιβόμαστε για το τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει το Συμβούλιο το Κοινοβούλιο και σας θυμίζω ότι εδώ πρόκειται για τραπεζική και χρηματοπιστωτική εποπτεία και οι τέσσερις συντονιστές των μεγάλων, πιο μεγάλων ομάδων ήταν, είπανε όταν το ΕΚΟΦΗΝ έκρινε ότι έκλεισε το θέμα ότι το Κοινοβούλιο είχε εξίσου δικαιώματα όπως και το Συμβούλιο. Δεν ήταν ε, θέση επί της ουσίας, ήταν θέση όσον αφορά τις αρμοδιότητες του Κοινοβουλίου. Υποστηρίζουμε λοιπόν απόλυτα αυτό που περιγράψατε. Εκτιμούμε σωστό το πρόγραμμα εργασίας αυτό, παρά το μεγάλο φόρτο εργασίας της Επιτροπής μας, αντέδρασε αποτελεσματικά στη χρηματοπιστωτική κατάσταση έχετε την πλήρη υποστήριξή μας. Αυτό ήθελα να σας πω. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Ζωζέ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Εγώ έρχομαι στο θέμα αυτό το οποίο έθεσε ο συντονιστής μου και πρέπει να πω ότι εγώ απογοητεύομαι από τη στάση του Συμβουλίου όταν προβλέπεται να είναι παρούσα η Υπουργό Οικονομικών και δεν έρχεται. Ήξερα ότι στις 26 και 27 που έγινε η συνάντηση με τα Εθνικά Κοινοβούλια χρειάστηκε να φύγει από την αίθουσα η κυρία Υπουργό, αλλά δεν καταλαβαίνω γιατί η Υφυπουργός δεν μπορούσε, ο Υφυπουργό δεν μπορούσε να είναι παρόν εκεί, ούτε σήμερα εδώ ενώπιον μας για να την αντικαταστήσει. Και αυτό είναι κάτι το οποίο έχει να κάνει με τη σχέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με το Συμβούλιο. Η πρώτη φορά που κάνω μια συνάντηση με το Συμβούλιο σε θέματα χρηματοοικονομικής εποπτείας ήταν η προηγούμενη εβδομάδα. Μέχρι τότε δεν υπήρξε καμία γνώση από τη δική μας πλευρά για τις προθέσεις του Συμβουλίου. Σε τέτοιες συνθήκες είναι πολύ δύσκολο να προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε τις θέσεις μας με το Συμβούλιο για να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε μία έγκριση σε πρώτη ανάγνωση του πακέτου που έχουμε ενώπιόν μας και εγώ Πιστεύω ότι πρέπει να κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες η πρόεδρος μας, ώστε το Κοινοβούλιο να κάνει ακουστή τη φωνή του. Είχαμε τέσσερις συνεδριάσεις για τα θέματα αυτά για την κρίση της Ελλάδος. Συζητούν όλοι οι συνάδελφοι. Θέλαμε σήμερα να έχουμε την Υπουργό Οικονομικών της Ισπανίας και φαίνεται σήμερα ότι πρέπει πάλι να μιλήσουμε μεταξύ μας. Μπορεί να είναι καλό αυτό για τη σωτηρία της ψυχής μας, αλλά εγώ νομίζω ότι η πρόεδρος πρέπει να επιμείνει για να έχουμε πιο καλές σχέσεις με το Συμβούλιο για τα θέματα αυτά. Ευχαριστώ. Η Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε και εγώ συμμερίζομαι την ε, απογοήτευση πολλών για την μη παρουσία της κυρίας Αλγάδο ανεξάρτητα από τους λόγους που την εμποδίσουν να είναι παρούσα μεταξύ μας ξέρω ότι θέλετε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη στιγμή για να συζητήσετε λιγάκι τον τρόπο συζητήσουμε για τον τρόπο με τον οποίο το Κοινοβούλιο μπορεί να υπησέλθει σε θέματα μακροοικονομικά, θέματα που πολλές φορές τα έχουμε αντιμετωπίσει στο παρελθόν σε κατάσταση κατεπήγοντος, να μπορούμε να τα αντιμετωπίζουμε με ένα πιο τακτικό τρόπο. Πρόκειται για το θέμα της Ελλάδος σήμερα, το οποίο μας εγκαλεί σε σχέση με την ικανότητα διαχείρισης κρίσεων από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά έχουμε και την ευθύνη που πρέπει να επομιστούμε σε φυσιολογικέ καταστάσει για την διαχείριση τη οικονομική πολιτική. Αν δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό σε φυσιολογικέ συνθήκε, τι θα κάνουμε σε περίπτωση κρίση. Εγώ νομίζω ότι θα πρέπει να εξετάσουμε και τι δύο αυτέ πτυχέ και αυτά που πρέπει να δούμε αύριο σε μακροοικονομικό επίπεδο. Δεν είναι μονάχα η δημιουργία μηχανισμών αντιμετώπισης κρίσεων, αλλά είναι και τα θέματα γενικότερα οικονομικής ευκυβερνησίας. Θα πρέπει να κάνουμε μία διάκριση μεταξύ των δύο αυτών πτυχών και σε επίπεδο νομοθετικό, γιατί κάποιοι από εμά είναι σε διαπραγματεύση με το Συμβούλιο σε ό,τι αφορά το πακέτο εποπτείας και πρέπει να τονίσουμε το πόσο σημαντικό είναι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αν θέλουμε τα κείμενα αυτά να διατηρήσουν κάποιες πτυχές συλλογικού ευρωπαϊκού συμφέροντος και να μην απλώς αριθμητικό άθεσμα των απόψεων των κρατών μελών. Και δεν θέλουμε, δεν πρέπει να μας αφήσουν, να μας αφήσουμε να μας παγιδεύσει η οριακή ημερομηνία 1η Ιουλίου 2010 που υποτίθεται πρέπει να έχει τελειώσει η εξέταση του πακέτου για να τεθεί σε εφαρμογή την 1η Ιανουαρίου του 2011. Για τα θέματα της εποπτείας έχουμε ζητήσει εδώ και πολύ καιρό να υπάρξει πρόοδο στα θέματα αυτά και ξέρουμε ότι το πακέτο αυτό δεν θα ξανανοίξει από τη στιγμή που θα εγκριθεί. Πρώτο περάσουν πολλά χρόνια. Λοιπόν, είναι καλύτερο να περιμένουμε λιγάκι και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να κάνει σωστά το έργο του για να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε ένα πακέτο το οποίο δεν είναι ένα συνονθήλευμα προτάσεων, αλλά ένα συνακτικό σύνολο που μπορεί να αντιμετωπίσει όλα αυτά τα προβλήματα που όλοι μας γνωρίζουμε. Για τα μακροοικονομικά θέματα. <clears throat> Αναφερθήκατε στην ομάδα εργασία υπό την ε, γίδα του κυρίου Φαν Ρόμπεϊ. Για το Συμβούλιο, εγώ νομίζω ότι είναι θετικό αυτό το νέο. Πιστεύω ότι ο πρόεδρος Φαν έχει σαφώς μια πρόθεση να αντιμετωπίσει με φιλόδοξο τρόπο τα προβλήματα της οικονομικής πολιτικής. Αλλά το θέμα είναι πώς έχει καθοριστεί η εντολή του, της ομάδας αυτής της εργασίας. Ο πρώτος Φανερόμπερι την τελευταία στιγμή έδωσε ουσιαστικά <clears throat> ένα ε, σκαμνάκι στην Κομισιόν για να παίζει και αυτή. Ενώ είχαν αποφασιστεί μεταξύ των δύο μεγάλων κρατών μελών να υπάρχει αυτή η δημιουργία της ομάδας αυτής της εργασίας, δεν είχε προβλεφθεί η παρουσία της Κομισιόν. Η Κομισιόν τελικά φαίνεται ότι της δόθηκε μια μικρή συμμετοχή. Και το ανακοινωθέν στο 10 Μαΐου θα αναφέρεται ακριβώς σε αυτή τη νέα μορφή. Τώρα, σε τι θα χρησιμεύσει αυτή η ομάδα εργασίας. Εγώ λέω δύο πράγματα. Καταρχήν αυτή η ομάδα εργασίας θα έχει ενδεχομένως την ε, <clears throat> εντολή του να προτείνει τροποποίησης της συνθήκης. Και εξάλλου ο πρόεδρος Γιούνκερ θα ξέρει πώς θα λειτουργήσει αυτή η ομάδα, αλλά μάλλον θα απαρτίζεται από υπουργού οικονομικών. Μα αυτό σημαίνει στην πράξη μια διακυβερνητική διάσκεψη. Και η συνθήκη της Λισαβόνας είναι σε αυτήν την περίπτωση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την ε, δυνατότητα να ζητήσει να συγκληθεί μια συνέλευση σε τέτοιες περιπτώσεις μεταρρύθμιση των συνδικών. Ξέρω την πρωτοβουλία που αναλάβατε να ζητήσετε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να συμμετάσχει στις εργασίες αυτής της ομάδας εργασίας. Αλλά αυτό πραγματικά το ελάχιστο ελάχιστο. Μήπως όμως θα ήταν καλύτερο να ζητήσουμε εμείς να εκπροσωπηθεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλύτερα και όχι μονάχα από ένα εκπρόσωπο μεταξύ 27 Υπουργών Οικονομικών. Νομίζω ότι πρέπει να ξεπεράσουμε <clears throat> αυτό το στάδιο και να σκεφτούμε για το πώς θέλουμε να παρεύουμε σε Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στα θέματα αυτά. Όταν τελειώσει αυτή η άσκηση, είτε είναι για την φυσιολογική διακυβέρνηση, είτε για τους μηχανισμούς κρίσης, αν αυτό μας οδηγεί σε κάποιες λογικές προτάσεις και συμπεράσματα, επί τη βάση των προτάσεων της Κομισιόν, <clears throat> θα καταλήξουμε σε κάποια νομοθετικά κείμενα. Και το Κοινοβούλιο φυσικά θα εμπλακεί στη διαδικασία. Ελπίζουμε λοιπόν θα μπορέσουν να προχωρήσουν τα πράγματα. Έχουμε μια προφορική ερώτηση η οποία είναι υπό εκπώνηση. Θα έχουμε τη δυνατότητα να συζητήσουμε με την Κομισιόν μέσω και εκθέσεων πρωτοβουλίε μετά από την ανακοίνωση τη 12η Μαου. Η πρότασή μου όμω και το έχω πρόθεσή μου και το έχω αναφέρει και σε άλλου συναδέλφου είναι <clears throat> πέραν του καθαρά θεσμικού ρόλου που έχουμε μέσω της νομοθετικής διαδικασίας και των εκθέσεων πρωτοβουλίας να προσπαθήσουμε να κάνουμε αυτό το οποίο θα θέλαμε να είχε κάνει ήδη το Συμβούλιο. Γιατί ο κίνδυνος τη ομάδα εργασία του κ. Φαν Ρόμπα όσο καλή και να είναι αυτή η ομάδα εργασία, όσο μεγάλη εμπειρογνωμοσύνη να έχουν και καλή θέληση, <clears throat> είναι ότι με τον τρόπο αυτό μπαίνουμε στο παιχνίδι μιας διακυβερνητική διαπραγμάτευση. Ενώ αυτό το οποίο χρειαζόμαστε είναι να μπορέσουμε να επανεύρουμε το συλλογικό ευρωπαϊκό συμφέρον και την ευρωπαϊκή προσθέμενη αξία. Γι' αυτό προτείνουμε εμείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να αναλάβουμε <clears throat> την πρωτοβουλία με τη δική μας ευθύνη να δημιουργήσουμε μια ομάδα σοφών η οποία εν παραλίλω θα εκπονήσει προτάσεις και αυτό θα μπορέσει να οδηγήσει σε μια συζήτηση, σε ένα διάλογο που να έχει ακαδημαϊκούς, οικονομολόγους, νομομαθείς, ώστε η συζήτηση να μην παραμείνει με <clears throat> μέσα σε ένα στενό διακυβερνητικό πλαίσιο. Αυτό είναι αυτό που βλέπω με την τωρινή σύνθεση αυτής της ομάδας εργασίας. Συγγνώμη που μακρηγορώ, επειδή όμως δεν είμαστε πολύ αριθμοί, νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να σας παρουσιάσω αυτή την πρόταση. Ευχαριστώ. Ε, Ευχαριστώ, Με χαρά πάντα σε ακούμε, γιατί ήσουν και πρόεδρος της Επιτροπής αυτής και πολλών άλλων. Ο Σφεν και μετά η Άννη, ο κύριος Χουντής, κάποιος άλλος που δεν έχει μπει στο κατάλογό μου, η Βίκη. Ωραία, Σφεν. Δεν είμαι σίγουρος. Τώρα ε, δεν επικεντρωνόμαστε τόσο πολύ στα ουσιώδη, αλλά στο ρόλο του Κοινοβουλίου στην όλη διαδικασία. Μια που έχουμε χρόνο καλό θα ήταν να δώσουμε έτσι μια δομή στη συζήτηση. για τα ουσιώδες του πράγματος. Έχουμε καλούς λόγους που μας οδηγούν στην σημερινή συζήτηση. Γιατί τουλάχιστον στα γερμανικά έψιλον άκουσα πολλά μπρος πίσω με τον ε, κύριο Λάγκιν, ο οποίος ήθελε να βγει η Ελλάδα από την Ευρωζώνη. Απ' την άλλη ακούσαμε άλλη θέση από άλλα μέλη του ΕΛΚ. Ακούστηκαν διάφορες απόψεις. Οπότε έχει νόημα αυτή η συζήτηση. Αλλά βέβαια νομίζω ότι κρίμα είναι που δεν, μπορούσαμε, δεν μπορέσαμε να προχωρήσουμε με το σχέδιο ψηφίσματος που ήδη είχαμε προετοιμάσει. Νομίζω ότι πολλά καλά επιχειρήματα ακούστηκαν, υπευλήθησαν τροπολογίες, ακούστηκαν πολλές απόψεις. Οπότε αν κάποιοι δεν είναι ικανοποιημένοι με ένα κομμάτι του, εντάξει να το συζητούσαμε. Αλλά τώρα έχουμε μείνει πίσω. Οπότε τώρα αν παραπονούμεθα ότι ο ρόλος του Κοινοβουλίου δεν θεωρείται όσο σημαντικός θα έπρεπε από το Συμβούλιο, ε, δεν θα έπρεπε να μας εκπλήσει αυτό, γιατί κάνουμε τόσες εβδομάδες δουλειά και μετά δεν μπορούμε να ψηφίσουμε το αποτέλεσμα της δουλειά μας. Οπότε πραγματικά εμένα με λυπεί αυτό. Και είναι κρίμα που δεν μπορέσαμε να προχωρήσουμε και να έχουμε μια ισχυρή θέση. Θα ήταν νομίζω δυνατόν να διαπραγματευτούμε λίγο περισσότερο ώστε να καταλήξουμε σε μια συμφωνία ε, μεταξύ των πιο φεντεραλιστικών ομάδων. Αλλά είναι κρίμα που έχουμε τώρα αυτό το εμπόδιο. Και θα ήθελα και την άποψη των υπολείπων. Δεν πήγε χαμένη η δουλειά μας τελικά. Θα επανέλθουμε σε κάποιο μεταγενέστερη χρονική στιγμή στο ψήφισμα. Δεν νομίζω ότι θα ήταν καλό αυτό. Αυτά για τη διαδικασία και για τα πιο ουσιώδη θα σας τα πω αργότερα. Ευχαριστώ. Όχι, δεν θυσιάσαμε τη δουλειά που κάναμε. Απλώς κάποιοι θεώρησαν ότι χρειάζεται περισσότερο χρόνος για να απαντήσουμε καλύτερα στο Συμβούλιο. Φαντάζομαι όμως ότι θα επανέλθουμε. Η κυρία Ποδηματά έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ε, συμπυκνώσατε με εξαιρετικό τρόπο τις ε, αποφάσεις που λήφθησαν το τελευταίο τριήμερο για την ενεργοποίηση του μηχανισμού στήριξης. Θέλω πρώτα απ' όλα να πω ότι προσπογράφω και συμφωνώ απολύτως και με την πρόταση της Περβάνς ε, για την ε, σύσταση μιας Επιτροπής Οφών στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που θα παρακολουθεί και θα συμβάλλει στις συζητήσεις που έχουν ξεκινήσει για την ενίσχυση της οικονομικής ε, ε, διακυβέρνησης και με την επισήμανση του ΣΒΕΝ. Και με αυτή την αφορμή ήθελα πάρα πολύ σύντομα να σας πω ε, μερικά στοιχεία για τη συμφωνία που επετεύθηκε την Κυριακή για την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων δηλαδή ανάμεσα στην Τρόικα και τις ελληνικές αρχές που κατέληξαν όπως γνωρίζετε στο πιο αυστηρό και σκληρό πρόγραμμα δημοσιονομικής ε, εξυγίανσης που έχει εφαρμοστεί ποτέ ε, στην Ευρώπη προκειμένου να ενεργοποιηθεί ο μηχανισμός στήριξης των 110 δισεκατομμυρίων ε, ευρώ. Το πρόγραμμα αυτό έχει τρεις πυλώνες. Ο ένας πυλώνας αφορά στη δημοσιονομική προσαρμογή, ο δεύτερος πυλώνας στις διαρθρωτικές αλλαγές που θα πρέπει να γίνουν για να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας και ο τρίτος αφορά σε ένα μηχανισμό στήριξης του τραπεζικού συστήματος. Ε, ο στόχος είναι το δημοσιονομικό έλλειμμα να μειωθεί κατά 6% του ΑΕΠ το 2010. Έχουν σημασία τα νούμερα, γι' αυτό επιμένω. Από 13,6% δηλαδή ε, με έτος βάσης το το 2009 ε, να φτάσει το 8,1% στο τέλος του χρόνου, 7,6% το 2011, 6,5% το 2012, 4,9% το 2013 και κάτω από 3%, δηλαδή 2,6% το 2014. Αυτή είναι η στόχη που αποτυπώνονται στο τριετές πρόγραμμα που συμφωνήθηκε ε, με την, με την Τρόικα. Ενώ σε ό,τι αφορά το δημόσιο χρέος προβλέπεται ότι θα αρχίσει να αποκλιμακώνεται από το 2013 και μετά. Είπα ότι πρόκειται για το πιο σκληρό και αυστηρό πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής που έχει εφαρμοστεί ποτέ ε, στην Ευρώπη. Ενδεικτικά σας λέω ε, ότι το πρόγραμμα, το πρόγραμμα προβλέπει ε, μείωση των αποδοχών στο δημόσιο τομέα, κατάργηση δύο μισθών, μείωση των συντάξεων, 8% ε, περαιτέρω μείωση των επιδομάτων για τους δημόσιους υπαλλήλους, ε, ουσιαστική αύξηση του συντελεστή φόρου προστιθέμενης αξίας από το 21% στο 23% και από το 10% στο 11%, αύξηση των ειδικών φόρων κατανάλωσης σε καύσιμα, τσιγάρα και ποτά, ε, νέο φορολογικό σύστημα και νέο ασφαλιστικό σύστημα σε ό,τι αφορά τις διαφορετικές αλλαγές. Θέλω επίσης να σημειώσω γιατί έχει τη σημασία ότι η εφαρμογή του προγράμματος θα παρακολουθείται όπως έχει ήδη ανακοινωθεί ανατρίμηνο από την Τρόικα και οι εκταμιεύσεις θα είναι συνάρτηση της επίτευξης κάθε φορά των στόχων που έχουν τεθεί. Και με αυτή την έννοια, και καταλήγω σε αυτό που κατά βάση θέλω να υπογραμμίσω, πρόκειται για ένα πάρα πολύ δύσκολο εγχείρημα, για ένα πολύ μεγάλο στίχημα, που όπως νομίζω ε, αγαπητοί συνάδελφοι, ότι όλοι και εμείς στην Ελλάδα και βεβαίω τα συμβαλόμενα μέρη του μηχανισμού ε, στήριξης αλλά και η Ευρωζώνη στο σύνολό της ε, έχουμε συμφέρον να προχωρήσει η υλοποίηση αυτού του προγράμματος όσο το δυνατόν πιο ομαλά με τις μικρότερες δυνατές ε, αναταράξεις, με τη μεγαλύτερη αποφασιστικότητα και με τις λιγότερες δυνατές διχογνωμίες και καθυστερήσεις, διότι διαπιστώσαμε όλοι το προηγούμενο διάστημα ότι οι καθυστερήσεις και οι διχογνωμίες πληρώθηκαν και εξακολουθούν να πληρώνονται ακριβά. Νομίζω λοιπόν ότι το Κοινοβούλιο, ε, για να συνδέσω με αυτά που έλεγε πριν και η Περβάνς, μπορεί και πρέπει να παίξει έναν αποφασιστικό ρόλο προς αυτή την κατεύθυνση. Τι εννοώ. Υπάρχουν ε, συμπεράσματα, διδάγματα που αντλούνται από την ελληνική κρίση. Η Επιτροπή μας έχει προχωρήσει σε μια σειρά από θετικές πρωτοβουλίες για να ε, εξάγουμε αυτά τα διδάγματα και αυτά τα συμπεράσματα. Ε, η ε, ελληνική κρίση, το ελληνικό δημοσιονομικό πρόβλημα έχει ασφαλώς μια βασική εθνική παράμετρο, ταυτοχρόνως όμως η δραματική επιδίωσή του, επιδίνωσή του τις τελευταίες εβδομάδες φέρνει στο προσκήνιο την ευρωπαϊκή διάσταση, τη διάσταση δηλαδή της έλλειψης αποφασιστικότητας και κοινών στόχων από την πλευρά της Ευρωζώνης και φέρνει επίσης στο προσκήνιο σε μια συγκυρία μάλιστα ιδιαίτερα ευτυχή γιατί όπως ε, είπε και η συζητάμε ε, το νέο εποπτικό πακέτο για το χρηματοπιστωτικό σύστημα τις ε, αδυναμίες που αφορούν στον έλεγχο και στην εποπτεία του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Επειδή λοιπόν βλέπουμε ότι ήδη υπάρχουν τα πρώτα σημάδια που απειλούν και άλλες χώρες της Ευρωζώνης Νομίζω ότι θα πρέπει ε, εμείς στο πλαίσιο της Επιτροπής μας αλλά και συνολικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, να δείξουμε μεγαλύτερη ε, αποφασιστικότητα και γενναιότητα σε ό,τι αφορά την εξαγωγή των συμπερασμάτων που θα πρέπει να βγουν για το θέμα της ενίσχυσης οικονομικής διακυβέρνησης και για την εποπτεία των αγορών και το δεύτερο, με το οποίο ολοκληρώνω, για να βοηθήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στην όσο το δυνατόν πιο ομαλή εφαρμογή των όσων συμφωνήθηκαν την προηγούμενη Κυριακή και για να είναι όσο το δυνατόν πιο ομαλή εφαρμογή αυτών που συμφωνήθηκαν την Κυριακή ε, θα πρέπει ε, οι Έλληνες πολίτες που καλούνται κατά βάση να σηκώσουν το μεγάλο βάρος αυτής ε, της προσπάθειας να έχουν μία αίσθηση ε, κατανόησης από την ε, πλευρά των υπολείπων ε, Ευρωπαίων εταίρων, από την πλευρά των άλλων ευρωπαϊκών πρωτευουσών και συμπαράστασης σε έναν εξαιρετικά δύσκολο δρόμο που υπάρχει μπροστά τους. Ευχαριστώ πολύ. πολύ, ο κύριος Χουντής. Αυτή ήταν στον, στον κατάλογο. Ο Ιμανουέλ θα ήθελε να επανέλθει και η κυρία Κράτσα τελευταία στη λίστα. Θέλει κανείς άλλος να μιλήσει πίσω τώρα και η Σόφια. Ο κύριος Χουντής έχει το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Το πρώτο μου σχόλιο έχει σχέση με τη διαδικασία και τα θεσμικά προβλήματα που έχει δημιουργήσει η κατάσταση έτσι όπως την περιγράψατε συνοπτικά και που αφορά καταρχήν την υπόθεση της Ελλάδας, αλλά όχι μόνο. Συμφωνώ με τις παρατηρήσεις που κάνετε σε σχέση με τον τρόπο αντιμετώπισης από την πλευρά του Συμβουλίου, της Επιτροπής μας και κατ' επέκταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Υπάρχει μια δεοντολογία, αλλά κατά τη γνώμη μου εγείρονται και θεσμικά ζητήματα, ακόμα και ζητήματα τήρησης της συνθήκης. Τι εννοώ με αυτό. Το πρόγραμμα το οποίο υπέγραψε και καλείται να εφαρμόσει η Ελλάδα με την Τρόικα προβληματίζει και την ελληνική πολιτική σκηνή αν πρόκειται για μια διεθνή συνθήκη η οποία ενδεχομένως περιορίζει την εθνική κυριαρχία. Αν πρόκειται για τέτοια συνθήκη, τότε η έστω και εκ των υστέρων συζήτηση που θα γίνει αύριο μεθαύριο στο Ελληνικό Κοινοβούλιο απαιτεί διαφορετικές πλειοψηφίες για να επικυρωθεί. Η δεύτερη πλευρά, αν είναι διεθνή συμφωνία αυτό, δηλαδή είναι συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με έναν εξωτερικό οργανισμό, στην προκειμένη περίπτωση του Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, τότε, τότε σύμφωνα με το άρθρο 218 της Συνθήκης έχει λόγο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι πρέπει και από αυτή την πλευρά να ειδωθεί το θέμα. Πολιτικά όμως, νομίζω κυρία Πρόεδρε, στο πλαίσιο της λογικής που αναπτύξατε ότι πρέπει να υπερασπιστούμε το ρόλο μας και τώρα και στις μελλοντικές διαπραγματεύσεις και επεξεργασία των συνδικών να ζητήσουμε σε κάθε περίπτωση, αυτή είναι η πρότασή μου, το πακέτο, η όλη συζήτηση, η όλη διαπραγμάτευση, η όλη συμφωνία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της ε, Κομισιόν και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου με την Ελλάδα να συζητηθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Για τους λόγους που προσπάθησα να εξηγήσω και ενδεχομένως και για λόγους πολιτικής δεοντολογίας είναι ένα κρίσιμο θέμα, δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, αφορά και άλλες χώρες. Είναι μια πρωτότυπη συμφωνία, δεν έχει ξαναγίνει τέτοιο πράγμα και επομένως κατά τη γνώμη μου και με βάση τις συνθήκες ε, ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ρόλο, έχει λόγο και πρέπει να τον υπερασπιστούμε. Εν γέννη, είμαι σύμφωνος με τις προτάσεις που διατύπωσαν οι ε, αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφισες που έχουν σχέση με το ότι πρέπει να διεκδικήσουμε ρόλο και στην ε, αναθεώρηση των συνθηκών και στους μηχανισμούς εποπτείας. Νομίζω ότι οι αποφασιστική θεσμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης με βάση και τους χειρισμούς της προηγούμενης περίοδου, τους χειρισμούς αυτή της περίοδου, θα πω δύο κουβέντες ακόμα, ε, και την εν γέννη πολιτική που ακολούθησαν, δεν συγκροτούν, δεν συγκεντρώνουν την απαραίτητη αξιοπιστία. Σίγουρα δεν είναι αξιόπιστη, ε, θα έλεγα, στους ε, πολίτες των ευρωπαϊκών χωρών. Ενδεχομένως να είναι μια αυστηρή κρίση, μπορώ να την τεκμηριώσω, δεν θα επεκταθώ περισσότερο σε αυτό. Η δεύτερη μου παρατήρηση έχει να κάνει με αυτόν τον μηχανισμό, με αυτή τη συμφωνία που συνήψε η Ελλάδα με την Τρόικα. Πρώτα απ' όλα, <clears throat> ακόμα δεν έχει απαντηθεί το ερώτημα κατά τη γνώμη μου, το οποίο δεν είναι απλό, τι δουλειά είχε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο σε ένα τέτοιο μηχανισμό στήριξης, ενώ υπήρχε η δυνατότητα, κατά την άποψή μου, σύμφωνα με το άρθρο 122 παράγραφος 2 της Συνθήκης, περί έκτακτης κατάστασης, η λύση να είναι σε κάθε περίπτωση ευρωπαϊκή. Δεν έχουν δοθεί, κατά τη γνώμη μου, πιστικές απαντήσεις, αλλά σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι αποτελεί για κομβικό σημείο η συμμετοχή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στα της Ευρωζώνης. Το δεύτερο, τα μέτρα που περιλαμβάνει ο μηχανισμός και τα οποία, όπως είπε και η συναδέλφισσα, είναι τα αυστηρότερα που έχουν ακουστεί όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, συνιστούν μονόπλευρες θυσίες, θα βαθύνουν την ύφεση στην Ελλάδα, δεν θα υπάρξει περιθώριο ή ελαχιστοποιούνται τα περιθώρια ανάπτυξης και κατόπιν τούτου στο τέλος θα είναι και αναποτελεσματικά και επομένως α, οι νέες δηλώσεις που κάνουν δυστυχώς ας πούμε ο κύριος Τρισέ υπενισόμενος ότι δεν φτάνουν αυτά τα μέτρα θα χρειαστούν και άλλα ίσως έχουν βάση αλλά από την άλλη άποψη δείχνουν ότι η Ελλάδα θα είναι για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα υπό την ασφικτική κυδαιμονία της Τρόικα αλλά σίγουρα τον πρώτο λόγο τον έχει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο αυτό επέβαλε τους όρους η Κεντρική Τράπεζα, αν παρακολουθήσατε προηγούμενη συζήτηση, δεν είχε δώσει απάντηση ποιο έχει τον πρώτο λόγο, ποιο βάζει του όρου. Ε, Επομένω, έχουμε μια χώρα τη Ευρωζώνης που θα είναι σε μια μακροχρόνια και δαιμονία εποπτεία του ε, εξωτερικού οργανισμού του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και αυτό σε κάθε περίπτωση δεν περιποιεί, δεν συγκροτεί ε, κύρος και ευθύνη σε όσου συγκροτούν την Ευρωζώνη και γενικά την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επαναλαμβάνω το ερώτημα, δεν έχει απαντηθεί. Και η τρίτη μου παρατήρηση είναι ότι με αφορμή την υπόθεση της Ελλάδας που τα γεγονότα και αυτών των ημερών η επίθεση στα, ε, στα ομόλογα της Πορτογαλίας, ενδεχομένως της Ισπανίας, δείχνει ότι δεν είναι μόνο ελληνικό πρόβλημα. Αποδεικνύονται διάφορες αγκυλώσεις και δομικά λάθη τα οποία δυστυχώς ε, δεν ε, βλέπω, δεν παρατηρώ την πρόθεση να συζητηθούν. Κατά τη γνώμη μου, έτσι όπως έχει συγκροτηθεί, έχει ιδρυθεί η ΟΝΕ και το ευρώ έχει δομικά λάθη. Το ευρώ δεν μπορεί να γίνει καλύτερο διότι δεν υπάρχει ισχυρός κοινοτικό προπολογισμό και δεν βλέπω πρόθεση να ενισχυροποιηθεί, δεν έχει εξασφαλιστεί η κινητικότητα της εργασίας και τρίτο και σημαντικό που πια είναι μπροστά μας, δεν υπάρχει μηχανισμός αντιμετώπισης της κρίσης, μηχανισμός δανεισμού έσχατης καταφυγής. Με με συνέπεια να έχουμε αυτά τα προβλήματα Προβλήματα έχουν και οι περισσότερες χώρες της ΟΝΕ, για να μην πω όλες, σε σχέση με το χρέος και τα ελλείμματα. Άρα ο προβληματισμός και η ενδεχόμενη συζήτηση για μεταρρύθμιση των συνθήκων πρέπει να ακουμπάει ή να θεραπεύει, αν είναι δυνατόν και αν υπάρχει τέτοια πρόθεση, τέτοια δομικά προβλήματα, διότι επαναλαμβάνω και τελειώνω εδώ για να μην σας κουράζω, είχαμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε, αν δεν θεραπευτούν αυτά, το φαινόμενο της Ελλάδας θα επεκταθεί ή και θα διευρυνθεί και σε άλλες χώρες και αυτό δεν, αυτή η παρατήρηση δεν οφείλεται σε κανένα είδο ελληνικό πατριωτισμό, ότι εν πάση περιπτώσει δεν φταίμε. Υπάρχουν προβλήματα στην ελληνική οικονομία, αλλά νομίζω ότι η βάση που ε, διόγκωσε αυτά τα προβλήματα που σήμερα εμφανίζονται στην Ελλάδα είναι ε, το πώς έχει θεσπιστεί το ευρώ και βεβαίως η αντιαναπτυξιακή και αναποτελεσματική λειτουργία του Συμφώνου Σταθερότητας. Δεν θέλω να σας κουράσω περισσότερο. Ευχαριστώ πολύ. Thank you very much. Εγώ ευχαριστώ. Η Βίκη Φόρτ έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Σημερίζομαι την απογοήτευση και των υπολείπων μελών που ακύρωσε την σημερινή ακρόαση Προεδρία. Καταλαβαίνω βέβαια ότι το να βρούμε έναν τρόπο να λύσουμε το πρόβλημα της Ελλάδας δεν είναι πολύ εύκολο. Βέβαια στις αγορές υπάρχει η ιδέα ότι θα βρεθεί μια ε, διεθνής λύση και αυτή κάπως νερώθηκε. Οπότε λίγο με ανησυχεί η σημερινή ακύρωση γιατί δεν νομίζω ότι ουδετεροποιείται έτσι αυτή η εντύπωση που επικρατεί. Καλωσορίζω βέβαια και τη συμμετοχή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και αυτό τονίζει πραγματικά τη σημασία που, έχει το να συνεργάζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση με μη ευρωπαϊκούς οργανισμούς. Αυτό που βλέπουμε στα μέσα μαζική ενημέρωση και στι εφημερίδε είναι το πώς έχει οδηγήσει η κρίση στην Ελλάδα σε μια πιο ευρεία ε, και επίγουσα, επίγον, ε, επίγουσα να κοινωνική κρίση. Και ε, χαίρομαι που μπορούμε να δούμε το τι λένε οι Έλληνες συνάδελφοι που είναι εδώ για το πώς έχει η κατάσταση επιτόπου. Ε, Γενικώ όμως ε, πρέπει να πω ότι αυτό δείχνει γιατί είναι σημαντικό οι χώρες αυτές με μεγάλα ελλείμματα όπως και το Ηνωμένο Βασίλειο να αναλάβουν αποφασιστική δράση για να τακτοποιήσουν τα δημόσια οικονομικά τους. Όχι απλώς για να αποκαταστήσουν την, ε, την εμπιστοσύνη από τι αγορές αλλά για να έχουν και την εμπιστοσύνη του κοινού, τη κοινή γνώμη. Όσο δηλαδή μα ψήφισαν σε αυτέ τι θέσει που είμαστε σήμερα. Ευχαριστώ. Ο Σβέν επανέρχεται. Μην να μακρηγορήσω όμως γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο. Πάρα πολύ σύντομα. Έρχομαι από το τμήμα της Γερμανίας που θα κάνει εκλογές την Κυριακή. Πρέπει να πω ότι δεν είμαι ιδιαίτερα ε, ικανοποιημένος από αυτά που έγιναν στη Γερμανία μετά από σαφείς δηλώσεις το Φεβρουάριο και το Μάρτιο ότι η Ευρώπη δεν θα άφηνε την ε, Ελλάδα αβοήθητη, υπήρχε ο χρόνος για σιωπηρές διαπραγματεύσεις. Αυτή ήταν η χρονική εποχή λοιπόν, όταν η βασική συμφωνία θα μπορούσε να είχε τύχει λεπτομεριακής διαπραγμάτευσης. Λόγω της ιδιαίτερης κατάστασης όμως στην χώρα μου, όπου είναι γνωστό ότι τα κόμματα τα οποία έχουν την εξουσία στο τμήμα αυτό της Γερμανία στη Βόρεια Ιρλανδία Βεσφαλία που παίζει και μεγάλο ρόλο στην πλειοψηφία στην Bundesrat στη δεύτερη Γερμανική Βουλή <clears throat> ήταν φανερό από τις δημοσκοπήσεις ότι δεν νιώθανε ιδιαίτερη άνεση με οποιαδήποτε βοήθεια προς την Ελλάδα και υπήρχε η διάχυτη ανάγκη να υπάρξει πιο στεναρή αντιμετώπιση των προβλημάτων. Αυτός είναι τελικά και ο αποχρόν λόγος, από την νομίζω, για τη στεναρή στάση που ακολούθησε η Γερμανία, η οποία δημιούργησε και περαιτέρω ανησυχίες και διαταραχές στις ε, αγορές και οδήγησε τα spread στα ύψη. Ο κύριος λόγος για όλα αυτά τα προβλήματα βέβαια, θέλω να το πω αυτό το πράγμα, ένας λόγος που δημιουργήθηκε από την ίδια την Ελλάδα. Και δεν συμφωνώ με αυτούς στο γερμανικό τύπο που είπαν ότι αυτό είναι ένα γενικευμένο πρόβλημα έλλειψης ισορροπίας στον ευρωπαϊκό χώρο. Όχι, υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα στην Ελλάδα. Δεν μπορεί κανείς να το, να το κρύψει αυτό. Υπάρχουν και άλλες χώρες στην Ευρώπη που έχουν πολύ υψηλό επίπεδο ε, χρέους και συγχρόνως μεγάλο έλλειμμα του προϋπολογισμού. Υπάρχουν μεγάλα βαθιά προβλήματα στην οικοδόμηση της Ευρωζώνης. Το έχουμε συζητήσει πολλές φορές υπήρξαν διαφορέ απόψεων για το πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτές τις ανισότητες και την έλλειψη ομοιόμορφης αντιαγωνιστικότητας. Νομίζω ότι η ελληνική κρίση καταδεικνύει ότι πρέπει να γίνει κάτι για να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα των ανισοτήτων μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η κλιμάκωση εξάλλου του προβλήματος οφείλεται στο γεγονός ότι το Συμβούλιο και η Γερμανία δεν έδωσε σαφή μηνύματα δεν ήταν μοναχά η γερμανική κυβέρνηση, ήταν η μεγαλύτερη, μεγαλύτερη κυκλοφορία εφημερίδα μας, η οποία ξεκίνησε μια μεγάλη εκστρατεία λέγοντας «Μη δώσετε πεντάρα στην, στην Ελλάδα», ακολουθώντας την άποψη αυτών των οικονομολόγων που λένε «Αφήστε τις αγορές μόνες τους, μην έχετε καμιά ρύθμιση στις χρηματαγορές» και δημιουργούσε αυτή την εντύπωση, την άποψη ότι θα πρέπει η αγορά να τιμωρεί αυτούς που κάνουν λάθη και μη βοηθάτε καθόλου αυτούς που δεν πάνε καλά. Εγώ δεν το είδα αυτό να υπάρχει πουθενά στην Ευρωπαϊκή Συνθήκη. Εγώ διαβάζω διαφορετικά την Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρά το γεγονό βέβαια ότι είναι σαφές πρέπει να γίνουν μεγάλες αλλαγές στην Ελλάδα, εκβάθρων αλλαγές. Και εγώ με την επίκριση του προγράμματος ότι είναι ένα πολύ σκληρό πρόγραμμα, αλλά πέραν αυτού θα πρέπει να αναφέρουμε ότι υπήρχε και πολλή ε, πλούτος ο οποίος βγήκε από το κύκλωμα λόγω πολιτι... πελατειακών, σχέσεων και πελατειακών πολιτικών που υποβοηθήθηκε και από δικές μας εταιρείες όπως η Siemens η οποία πλήρωσε 100 εκατομμύρια σε μίζες και τα χρήματα αυτά δεν εμφανίστηκαν ποτέ. Και είμαστε και ένας από τους μεγαλύτερους εξαγωγείς όπλων προς την Ελλάδα. Αυτά τα χρήματα δεν θα επανέλθουν. Εγώ βέβαια επικρίνω το πρόγραμμα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου γιατί στα θέματα του πλούτου που είναι η άλλη πλευρά του χρέους, δεν κάνει τίποτα αυτό το πρόγραμμα για τη δημιουργία πλούτου. Πού λοιπόν βλέπετε να υπάρχει η επαναφορά του πλούτου από τους Έλληνες που το έχουν αποκομίσει αυτό το πλούτο με πελατειακές σχέσεις και με διαφθορά, πού θα μπορέσει, πώς θα μπορέσει να ανακτήσει αυτό η Ελλάδα και η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτά τα χρήματα για να καλύψει το χρέος και τις πραγματικές ανάγκες της Ελλάδος. Και αυτό είναι η βασική επίκριση ότι το πιο ασθενέ τμήμα του πληθυσμού είναι αυτό το οποίο πιέζεται ακόμα περισσότερο μέσα στο προγράμμα του Διεθνού Νομισματικού Ταμείου. Ο Χωσέ, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Εγώ πιστεύω ότι αυτή η συζήτηση θα την έχουμε και πάλι με τον αρμόδιο επίτροπο τον κύριο Μπαρνιέ. Σήμερα και χθες και σήμερα είναι μια σημαντική ημερομηνία. Ίσως γιατί για πρώτη φορά θα δούμε πώς μπορεί να λειτουργήσει το ευρώ σε δύσκολες συνθήκες. Γιατί έχουμε ζήσει 10 χρόνια με το ευρώ σε εύκολες συνθήκες. Αυτό δεν ήταν πρόβλημα. Αυτό το οποίο έγινε με την Ελλάδα είναι αυτό το οποίο έπρεπε να γίνει. Κάτι έπρεπε να κάνουμε γιατί στην αντίθετη περίπτωση θα, είχαμε δεχθεί, θα είχε δεχτεί η Ελλάδα ένα πάρα πολύ σοβαρό κτύπημα και η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Οικονομική και Νομισματική Ένωση επίσης και επίση και οι τράπεζες που είχαν τα ευρω... Ε, τα ελληνικά ομόλογα θα είχαν μεγάλα προβλήματα, θα ήταν κάτι αντίστοιχο με την αγορά των ομολόγων subprime στις Πολιτείες η κρίση που θα προξενούν Ό,τι έχει γίνει όμως έγινε <clears throat> καθυστερημένα, αυτό είναι σαφές. Ξέρουμε όλοι πώς αντέδρασαν οι αγορές κατά τη διάρκεια αυτής της κρίσης. Έγινε επίσης με λανθασμένο τρόπο γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα δυσβάστακτο, αβάστακτο χρηματοοικονομικό βάρος για μια χώρα που δεν μπορεί να το σηκώσει ένα βάρος που θα οδηγήσει σε σημαντική μείωση του ΑΕΠ της χώρας αυτής και θα είναι επομένως ακόμα πιο δύσκολο να μπορέσουν να, μειώσουν, να μειώσει η Ελλάδα το δημόσιο χρέος της. Αν είναι επαρκές ή όχι αυτό το πρόγραμμα θα το δείξει ο χρόνος, αλλά σχεδόν όλοι οι σχολιαστές και το δείχνει και η αντίδραση της αγοράς ότι δεν θα είναι επαρκές αυτό το πρόγραμμα και θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε εν καιρό πιο δραστικές λύσεις ή την ε, αναδιάρθρωση του χρέους της Ελλάδος ή την έξοδο της από τη ζώνη του ευρώ. Αλλά αυτό το οποίο θέλω να συζητήσω με το Συμβούλιο και πρέπει να συζητήσουμε και με την Κομισιόν είναι άλλα θέματα. Στα θέματα της οικονομικής και νομισματικής πολιτικής η δράση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ήταν σπασμωδική. Οι πρώτες δηλώσεις ήταν ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δεν πρέπει να παρέμβει σε ένα θέμα που είναι θέμα εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ζώνης του ευρώ. Στη συνέχεια όμως όταν συζητήθηκε η δυνατότητα να υπάρξει μια κοινή έκδοση ε, ομολόγων από τις χώρες της ζώνης του ευρώ που θα μείωνε το οικονομικό βάρος της Ελλάδος, τότε ελέγχθη, <clears throat> όπως είπε και ο Γκίγκολτ, ότι οι αγορές πρέπει να τιμωρήσουν τους κακούς μαθητές. Αυτούς οι οποίοι δεν έκαναν σωστά το ρόλο του και φυσικά αυτό δεν αφορούσε τους ε, χρηματοπιστωτικούς φορείς που έπαιξαν μεγάλο ρόλο στην κρίση και τους οποίους τους διασώσαμε με τα βαΐα και κλάδων και μεγάλης δαπάνης. Η κρίση έδειξε τις ε, ελλείψεις της ε, παρακολούθησης σε ό,τι αφορά τα στατιστικά στοιχεία της Ελλάδος. Είναι γεγονός ότι το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης δεν λειτουργεί καλά. Ήδη από το 2005 έχω ζητήσει να αναθεωρηθεί αυτό το Σύμφωνο Σταθερότητας τόνιζα ότι είναι απαραίτητο να ενισχύσουμε αυτό το σύμφωνο σταθερότητα, αλλά μέχρι στιγμή όπω έχει δεν λειτουργεί. Να σα δώσω ένα παράδειγμα. Στο 2007 στο Ηνωμένο Βασίλειο, μέσα σε οικονομική ανάπτυξη και με ένα τεράστιο χρηματοπιστωτικό τομέα, το Ηνωμένο Βασίλειο είχε ένα έλλειμμα 13%. Επομένως βλέπετε ότι δεν λειτουργούν τα πράγματα τόσο εύκολα. Η τελική δυνατότητα διάσωσης είναι η οικονομική ε, παροχή πόρων για να μην ε, χρεοκοπήσει μια χώρα. Ούτε και αυτό λειτουργεί. Με την Ελλάδα αυτή τη στιγμή, αν μπορέσει η Ελλάδα να βγει από αυτή τη μαύρη τρύπα και καταφέρει να επιτύχει επαρκή, ε, επαρκή ρυθμό ανάπτυξη, όλα αυτά τα μέτρα που παίρνουμε τώρα δεν πρόκειται να βοηθήσουν καθόλου και θα ξανάρθουμε στην ίδια κατάσταση. Γι' αυτό σα λέω και πάλι το να θέσουμε ένα οικονομικό βάρος της τάξης του 5% που είναι αυτό το οποίο αναφέρεται, νομίζω ότι αυτό δεν είναι η καλύτερη λύση. Thank you. Uh, κυρία Κράτσα. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω και σας προσωπικά και τα μέλη της Επιτροπής μας για την προσοχή που έχετε δείξει στη ελληνική περίπτωση και το χρόνο και τις συνεδριάσεις που έχουμε αφιερώσει. Θα ευχαριστήσω για την κατανόηση και την αλληλεγγύη, άλλοτε περισσότερο, άλλοτε λιγότερο βέβαια. Ε, πρέπει βέβαια να ομολογήσω ότι είναι και μια δύσκολη ελληνική περίπτωση, γιατί το ελληνικό πρόβλημα έχει βαθιές ρίζες. Αποδεικνύεται ότι το αναπτυξιακό μοντέλο που ακολουθήσαμε δεν ήταν επιτυχές ε, και έχουν ακυρωθεί πολλές δυνατότητες που είχε χώρα και ο δημιουργικός ε, χαρακτήρας των κατοίκων, των Ελλήνων και φυσικά οι παρεμβάσεις που έγιναν και οι δυνατότητες που έδιναν τα διαφορετικά ταμεία. Αυτό που θέλω να τονίσω σήμερα είναι την ανάγκη εμπλοκής των κοινοβουλίων, του ευρωπαϊκού, του ελληνικού φυσικά και των εθνικών κοινοβουλίων και στη διαχείριση αυτής της κρίσης και στην ε, ε, ε, προσπάθεια για μια επιτυχέστερη οικονομική διακυβέρνηση στην Ευρώπη. Δεν μπορεί τα κοινοβούλια να είναι εκτός αυτής της ε, υπόθεσης. Διότι εδώ αυτό που λείπει δεν είναι μόνο οι κατάλληλοι θεσμοί, έτσι λειτουργήσε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μετά από κάθε κρίση αποδεικνυόταν ότι οι θεσμοί δεν ήταν αρκετοί και τους ενισχύαμε, τους αλλάζαμε, τους εμπλουτίζαμε. Εδώ όμως είναι και θέματα παρακολούθησης, θέματα αναπτυξιακής πορείας. Αφού κάθε τρεις μήνες θα αξιολογείται το ελληνικό πρόγραμμα, είναι πολύ σημαντικό, αυτό θέλω να τονίσω σήμερα, να έχει άποψη το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το Ελληνικό Κοινοβούλιο πρέπει να αποκτήσει μια ουσιαστική εμπλοκή και όχι τυπικά έγκριση προϋπολογισμών και τυπικά έγκριση εκτέλεσης των προϋπολογισμών όπως γίνεται μέχρι τώρα. Πρέπει να, ε, ε, ε, να αποκτήσει μια δημο, κουλτούρα δημοσιονομικού ελέγχου και τέτοιων θεσμών αλλά και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να παρακολουθεί στα, ε, τα προγράμματα αξιολόγηση που θα κάνει η Κομισιόν, διότι ο κίνδυνος στην Ελλάδα σήμερα είναι να μην μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη, άρα δημιουργία πηγές εσόδων. Μόνο με, με, μέσα τα οποία μέχρι τώρα ε, φαίνονται σαν κύρια μέσα, ε, είναι ένα πρόβλημα το οποίο δεν θα δώσει πόρους, ευκαιρίες δημιουργία ελπίδα για δημιουργία επιχειρήσεων, δημιουργία επενδύσεων, θέσεων εργασία. Λοιπόν, ο κίνδυνο είναι σήμερα η οικονομική και κοινωνική ύφεση και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να έχει άποψη διότι πρέπει να επισημάνουμε την ανάγκη παράλληλης αναπτυξιακού σοκ στην Ελλάδα μαζί με τα ε, ε, μέτρα δημοσιονομικής πειθαρχίας. Από την άλλη μεριά υπάρχει ανάγκη για διαδραστικές αλλαγές, αλλαγές στις οποίες ε, σχεδιάσαμε, υπολογίσαμε και δεν ε, κάναμε λόγω πολιτικού κόστους και μη πολιτική συνένεση τα προηγούμενα χρόνια και όλα αυτά που ξέρουμε πια ότι είναι παθογένειες και τα ομολογούμε σε ελληνικό επίπεδο και τα συζητούμε πια σε ευρωπαϊκό επίπεδο, δεν είναι πια ένα εθνικό μας μόνο θέμα, καλό είναι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να παρακολουθήσει και να... Ε, ε, ε, βοηθήσει την αλλαγή αυτού του αναπτυξιακού μοντέλου στη χώρα μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Ε, και βέβαια, ε, με συγχωρείτε κύριε Πρόεδρε, το άλλο θέμα βέβαια είναι νομικό. Και πιστεύω ότι πρέπει να έχουμε νομική άποψη και από την Ελληνική Βουλή, γι' αυτό που ο κύριος Κουντής, αν θα πρέπει να θεωρηθεί μια συμφωνία με διεθνή οργανισμό ή μια εσωτερική υπόθεση το πρόγραμμα αυτό ο, της Ελλάδος ή αν θα πρέπει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να έχει μια άποψη σαν μια ε, ε, συνθήκη με έναν ε, διεθνή οργανισμό όπως είναι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Νομίζω ότι χρειαζόμαστε μια συμβουλή νομική. Ευχαριστώ. Αρχίζω να αισθάνομαι ότι θα πρέπει να ζητήσουμε τη γνώμη των νομικών υπηρεσιών μας για μερικά θέματα που ήδη ετέθησαν. Ο Ούντο έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Δεν ήθελα να πω κάτι για την Ελλάδα, γιατί υπήρξαν πολλοί ομιλητέ προηγουμένω από μένα που αναφέρθηκαν στο θέμα αυτό. Θέλω να κάνω μονάχα μια παρατήρηση για αυτά που είπε ο Χωσέ Μανουέλ για την ε, ζώνη του ευρώ. Νομίζω ότι είπε κάτι το οποίο δεν νομίζω ότι έχει νόημα. Είπε ότι αν υπάρξει μια χώρα η οποία θα μείνει αβοήθητη, θα, ιδίως άμα βγει από τη ζώνη του ευρώ, τα, τα χρέη της θα εκραγούν όταν υποτιμηθεί σε σχέση με το ευρώ και έτσι κι αλλιώς οι κερδοσκόποι θα χτυπήσουν την επόμενη χώρα. Αυτό το οποίο φαίνεται σαφώς είναι ότι δεν έχουμε καθόλου μέτρα που θα εξασφαλίσουν καλύτερο συντονισμό στον οικονομικό χώρο στην Ευρώπη και επίση για τους κερδόσκόπου για τις ε, επενδυτικές τράπεζες θα πρέπει να υπάρξουν μέτρα και σε εθνικό επίπεδο και σε ε, ευρωπαϊκό επίπεδο και ιδίω σε ό,τι αφορά τη χρήση των παραγωγών. Εγώ συγκεντρώνω την προσοχή μου στο Συμβούλιο τώρα. Γιατί πιστεύω ότι αυτό το οποίο έχει παρουσιάσει το Συμβούλιο ως διαχείριση κρίσεως ήταν ολέθριο. Λόγω της καθυστέρησης τα πράγματα κλιμακωθήκανε, κερδοσκοπία αυξήθηκε και δυστυχώς πρέπει να πω στον κύριο Γκίγκολτ, δυστυχώς αυτό ήταν και κάτι στο οποίο οφείλεται και στην έλλειψη, στην απραξία της γερμανικής κυβέρνησης. Έχουμε όμως τώρα ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα ενώπιόν μας και πρέπει να διαπιστώσουμε ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο έχει προτεραιότητα ως πιστωτής, μετά θα έρθουν οι κερδοσκόποι και μετά τα κρατη τα οποία θα δώσουν διμερή βοήθεια. Αυτό δεν είναι πάρα πολύ άνετη θέση για τα κράτη-μέλη. Και αυτό είναι το αποτέλεσμα των ε, αμφιταλαντεύσεών τους και της μη αποφασισμένης πολιτικής που ακολούθησαν. Και εγώ ενδιαφέρομαι πολύ να ακούσω τι θα μας πει στις 12 Μαΐου ο Όλη Ρέν όταν παρουσιάσει τις δικές προτάσεις, προτάσεις της Κομισιόν. Αν προτείνει η Κομισιόν να δημιουργήσουμε ένα ευρωπαϊκό μηχανισμό αντιμετώπισης κρίσης που είναι κάτι περισσότερο από ένα μηχανισμό διμερούς χαρακτήρα μεταξύ κρατών μελών, εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να το υποστηρίξουμε. Πρέπει να έχουμε μια ευρωπαϊκή απάντηση σε τέτοιου είδους κρίσεις και όχι μονάχα μια, ε, ευρω... λύση σε διμερές επίπεδο που με εργόδη τηλεφωνήματα μεταξύ πρωτευουσών δημιουργείται μετά από μεγάλη καθυστέρηση. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι λοιπόν στο επόμενο κύμα κερδοσκοπία το οποίο μπορεί να χτυπήσει άλλε χώρε. Θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι να δώσουμε μια έγκαιρη και αποτελεσματική απάντηση. Ευχαριστώ. Κύριο Κλούτ. Ευχαριστώ. Εγώ δεν άκουσα κάποιον Έλληνα συνάδελφο ο οποίος να πει να διαφυσβητήσει ότι υπήρχαν προβλήματα στην Ελλάδα και ότι αυτά τα προβλήματα είναι το αίτιο της κρίσης. Αλλά θέλω να συνεχίσω αυτά που είπε ο Νίκος Χούντης. Κατά την άποψή μου, δεν πρόκειται μονάχα για ελληνικά αίτια για την κρίση αυτή. Και είδατε τα προβλήματα με την Πορτογαλία όταν υποβαθμίστηκε η επιστολιπτική του ικανότητα όπως και της Ισπανίας, βλέπετε ότι εδώ υπάρχει και κάποιος ευρύτερος λόγος. Θα ήταν χρήσιμο λοιπόν, θα ήταν πολύ λογικό να μην ασχοληθούμε αποκλειστικά μονάχα με τα εσωτερικά προβλήματα και να εστιάσουμε σε αυτά και μόνο. Πιστεύω ότι και η, η γερμανική κυβέρνηση είχε ζητήσει να αφαιρεθεί και το δικαίωμα ψήφου για τα κράτη-μέλη τα οποία παραβιάζουν το Σύμφωνο σταθερότητα. Αυτό νομίζω ότι ήταν μια παράλογη πρόταση, αλλά ήδη φαίνεται και από το γεγονός ότι η κρίση ξεπερνάει μοναχά την Ελλάδα και είναι μια γενικότερη κρίση. Χρειάζεται λοιπόν να έχουμε και μια συζήτηση αυτού του θέματος στα πλαίσια της Στατηγικής Ευρωπαϊκής Ένωσης 2020. Αυτό είναι μια προέκταση σε κάποιο βαθμό της στρατηγικής της Λισαβόνας, αλλά θα πρέπει να δούμε κατά πόσο αυτή η στρατηγική η οποία αφορά αποκλειστικά το στόχο της ανταγωνιστικότητος και δεν κοιτάζει καθόλου τις ρίζες του κακού για την Ελλάδα, δεν ξέρω αν θα είναι υποφελής με τέτοια στρατηγική. Νομίζω ότι αυτό το οποίο βλέπουμε στην περίπτωση της Ελλάδος είναι ότι αν είχαμε ακολουθήσει πλήρως αυτή τη στρατηγική που θα είχε οδηγήσει σε πλήρη αποκρατικοποίηση, αυτό θα είχε οδηγήσει σε ακόμα μεγαλύτερη αδυναμία του συστήματος. Δεν θέλω τώρα να καταδαπανίσω το χρόνο για τα θέματα αυτά. Έχουμε πάντως οικονομικούς δείκτες που δείχνουν ότι πολλές φορές η, η οικονομία δεν μπορεί να λειτουργήσει λόγω δεν μπορεί να λειτουργήσει ακριβώς λόγω των μεταφορών πιστώσεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάση περιπτώσει, δεν πρέπει εμείς να εστιάσουμε την προσοχή μας αποκλειστικά στην Ελλάδα. Χρειάζεται μια ευρύτερη ανάλυση μέσα στο πλαίσιο και αυτής της αναδιατύπωσης της στρατηγικής για το 2020. Και χρειαζόμαστε και μια ευρύτερη αντιμετώπιση της ε, οικονομικής πολιτικής της ζώνη του ευρώ μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Υπάρχουν κάποιοι ακόμα που περιμένουν. Αντώνη και Σόφη, μετά ο Λίαμ και αν έχουμε χρόνο θα επανελθεί Άννη στο τέλος. Αλλά πρέπει να απαντήσουμε σε όλα αυτά. Ο Άντωνη έχει το λόγο. Αντώνιο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε και εγώ θα ήθελα να είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε με την κυρία Σαλγκάδο Καταλαβαίνω ότι είναι ένα πρόβλημα χρονοδιαγράμματος, ελπίζω στο μέλλον θα μπορέσουμε να το επιλύσουμε, αλλά αυτό δείχνει και τα προβλήματα λειτουργίας που έχουμε σε πραγματικό χρόνο. Μετά από τη συνθήκη τη Λισαβόνας θα ήταν χρήσιμο να κατανοήσουμε ότι έχουμε και νέου συνομιλητές για τα θέματα της ε, οικονομικής διακυβέρνησης, όπως ο πρόεδρος του Συμβουλίου και ο επικεφαλής του, της θα πρέπει λοιπόν να συμμετάσχουν όλοι αυτοί πιο ενεργά σε αυτή τη διαδικασία. Παίρναμε μια κρίση, διατρέχουμε μια κρίση και αυτή η κρίση δείχνει ότι δεν μπορούμε να διατηρήσουμε το status quo, θα πρέπει να επιφέρουμε θεμελιώδεις αλλαγές. Δεν είναι θέμα του ποιοι είναι καλοί και ποιοι είναι κακοί. Με τις μομφές και τις επιρρήψεις κατηγοριών δεν μπορούμε να επιλύσουμε τα προβλήματα. Θα πρέπει να δούμε με ποιο τρόπο μπορούμε να ξεφύγουμε από αυτή την κρίση. φαίνεται από την κρίση τι θέλουμε να τροποποιήσουμε. Θέλουμε να διατηρήσουμε την εσωτερική αγορά και το ενιαίο νόμισμα ή θεωρούν κάποιοι ότι τα προβλήματα αυτά θα επιληθούν καλύτερα αν αποδομήσουμε αυτά τα οποία είχαμε οικοδομήσει, να υπάρξει δηλαδή η κάθε χώρα να προστατευτεί πίσω από τα δικά της σύνορα και να προσπαθήσει να βρει έναν δρόμο μόνη της. Επομένω, αυτό το οποίο τίθεται αυτή τη στιγμή να είναι το αν η Ευρωσόνη είναι σε θέση να αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα στο σύνολό τη. Δεν είναι αποκλειστικά ένα ελληνικό πρόβλημα, είναι ένα πρόβλημα που αφορά όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και αφορά και το μέλλον τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Προφανώ υπήρξαν προβλήματα δυσλειτουργιών. Είναι σαφέ ότι υπήρξαν μεγάλε ελλείψεις σε ό,τι αφορά τη λειτουργία τη Οικονομική και Νομισματικής Ένωση. Και αυτό που βλέπουμε και τώρα είναι ότι δεν μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε επαρκώς σε πραγματικό χρόνο. Είναι πρόβλημα ευκυβενησίας. Προφανώς είναι σαφής ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας σε όλη αυτή τη διαδικασία, αλλά παρόλα αυτά το πρόβλημα είναι ότι δεν μπορούμε να έχουμε μοναχά μια νομισματική πολιτική αν τα κράτη δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν τις αγορές, Πώς μπορούμε να θεωρούμε ότι έχουμε κάποιες πολιτικές λογικές αντιμετώπισης των κίνδυνων. Σε ό,τι αφορά τώρα την βοήθεια προς την Ελλάδα, θα πρέπει να αναφέρουμε ποιοι είναι οι μηχανισμοί, ποιοι είναι οι στόχοι, ποιοι είναι οι έλεγχοι που πρέπει να τη συνοδεύουν και ποιε είναι και οι συνέπειε που θα προκύψουν σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πιστεύω πρέπει να προκύψουν και κάποιε συνέπειε σε ευρωπαϊκό επίπεδο, γιατί ο στόχο μα θα πρέπει να είναι να έχουμε μια μεγαλύτερη οικονομική ολοκλήρωση και όχι μονάχα να παρέχουμε βοήθειες. Το ερώτημα είναι βέβαια πιο βαθύ. Αν συνεχίσουμε να έχουμε ανισότητες μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, λόγω έλλειψης ευκυβερνησίας, τα προβλήματα αυτά θα οξυνθούν. Γι' αυτό χρειάζεται και μια πιο διαφροτική αντιμετώπιση στο πώς θα εξασφαλίσουμε την οικονομική πολιτική και τη διακυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση Υπάρχουν προβλήματα που έχουν να κάνουν με τον προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι και νομοθετικά θέματα και σε όλα αυτά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να έχει κάποιο λόγο για αυτά. Δεν μπορούν λοιπόν να ληφθούν αποφάσει σε αυτά τα επίπεδα χωρί την ενεργή συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και γι' αυτό υποστηρίζω αυτά που είπε και η Πρόεδρό μα, ότι το Κοινοβούλιο θα πρέπει να συμμετέχει πλήρω στη διαδικασία αυτή. Εφόσον διακυβεύεται το μέλλον τη Ευρωπαϊκή Ένωση, θα πρέπει να είμαστε παρόντε. Thank you, Sophie. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Επόδεινο το ξύπνημα αυτό και για την Ελλάδα και για την Ευρώπη. Γιατί δεν δείχνει μόνο τα προβλήματα της Ελλάδας, αλλά δείχνει και τις αδυναμίες τις εσωτερικές της Ευρωζώνης και καταδεικνύει και κάτι που το, το λένε κάποιοι εδώ και καιρό, ότι η νομισματική ένωση χρειάζεται και πολιτική ένωση. Αλλιώ είναι αδύνατο να δράσει, να αποφασίσει, να παρέμβει. Ελπίζω τώρα να τα καταφέρουμε. Να δώσουμε στην ε, Νομισματική Ένωση και τις απαραίτητες δομές για τη λήψη αποφάσεων. Τώρα, για την Ελλάδα. Να προσθέσω ότι είναι μια χώρα την οποία αγαπώ πολύ, οπότε δυστυχώς λυπάμαι και την κατάσταση. Ξέρω ότι η, κοινή γνώμη και σε άλλα κρατημέλια και στην Ελλάδα γίνεται όλο και πιο επιθετική και αν δούμε την, την Ελλάδα μόνη τη, καταλαβαίνω ότι οι άνθρωποι λένε ότι ναι, είναι πάρα πολύ σκληρά τα μέτρα, αλλά είναι και η ευθύνη των πολιτικών να εξηγήσουν ότι τα μέτρα αυτά δεν είναι α, σκληρά λόγω τη Ευρωπαϊκή Ένωση ή του, του Διεθνού Νομισματικού Ταμείου, αλλά λόγω των αλλαγών που έπρεπε να έχουν γίνει. Αν είχαν γίνει οι αλλαγέ πιο νωρί, δεν θα ήταν τόσο επώδυνα τα μέτρα τώρα. Επίση, απ' την άλλη, αποστασιοποιούμε λίγο από δηλώσει που γίνονται και σε εθνικό επίπεδο και στη δική μου χώρα και σε άλλες όπου ε, γίνεται έτσι μια γελιοποίηση κάποιων κρατών μελών, ε, δίνονται μόνο στερεότυπα, κάποια κράτη-μέλη θεωρούνται ε, υποδέστερα άλλων, αυτά είναι ιδίες. Σε αυτή τη φάση αυτό που πρέπει να γίνει είναι η... όλοι οι πολιτικοί να δώσουν υποστήριξη στην ελληνική κυβέρνηση, γιατί αυτό χρειάζεται έτσι ώστε να μπορέσει να εφαρμόσει αυτά τα μέτρα. Οπότε άκουσα τη συζήτηση και θα ήθελα και εγώ να ζητήσω στους συναδέλφους να αποφύγουν να σχολιάζουν ε, τις εθνικές πολιτικές, τις πολιτικές Ελλάδας. Τώρα, για τα μέτρα και το σχετικό πακέτο. Έλλειμμα και χρέος. Πρέπει να απαλληφθούν μέσω ε, ε, μειώσεων στον προπολογισμό. Από την άλλη, αυτό που λείπει είναι προτάσεις για οικονομική ανάπτυξη. Γιατί αυτό είναι η άλλη πλευρά του νομίσματος. Και τέλος, Πρόεδρε, να επαναλάβω αυτό που είπα και στην ακρόαση πριν από κανένα μήνα περίπου αυτή η κατάσταση όντως ζητά μια έτσι κοινοβουλευτική ε, ομοφωνία. Δεν μιλούμε μόνο για την Ελλάδα, μιλούμε για ένα σύστημα που δεν λειτουργεί καλά. Ξέρουμε ότι υπάρχουν και άλλα κράτη-μέλη που έχουν προβλήματα, όπου έχουν ε, εφαρμοστεί μέθοδοι που μπορεί να μην είναι πλήρως συμμορφούμενες με τους κανόνες και πρέπει να δούμε αν, όχι μόνο κατά πόσο έχουν γίνει λάθη, αλλά και πώς λειτουργεί τελικά το σύστημα και ποιος είναι ο ρόλος των κρατών μελών, πώς λειτουργεί το σύμφωνο σταθερότητας, η Κομισιόν και η Eurostat. Έχουν επαρκή εξουσία. Από ό,τι φαίνεται όχι. Έχουν χρησιμοποιήσει τις αρμοδιότητες του σωστά. Τι λείπει, γιατί λείπει, τι έχει γίνει μέχρι τώρα, πώς είναι δυνατόν Εάν χρόνια τώρα ξέρουμε ότι τα στατιστικά στοιχεία δεν ήταν σωστά, να μην έγινε τίποτα, να μην υπήρξε διορθωτικό μέτρο, πώς είναι δυνατόν αυτό. Και Εάν προσπαθούμε να κάνουμε ε, κοινοβουλευτικές έρευνες για την ε, τραπεζική κρίση, η νομισματική κρίση νομίζω αξίζει μία τέτοια διερεύνηση. Ίσως να, οδηγηθεί, να οδηγηθούμε και σε συμπεράσματα που να είναι ε, χρήσιμα και για, την, για το μέλλον του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Δέκα λεπτά έχουμε πριν έρθει ο κύριος Μπαρνιέ. Ο κύριος Βαγκόκ, ο Ζαν που είπε ότι θέλει να επανέλθει και μετά η Άννη. Ο Λίαμ. Ευχαριστώ. Εγώ ανήκω στην οικογένεια των φεντεραλιστών και είμαστε ικανοποιημένοι από το πρόγραμμα υποστήριξης προς την Ελλάδα, αν και θεωρώ ότι το 5% είναι κάπως ψηλό σαν νούμερο αλλά αν η Κεντρική Τράπεζα είχε κάνει όπως η Αμερικάνικη Κεντρική Τράπεζα, η Βρετανική Κεντρική Τράπεζα έκαναν, δηλαδή αν είχε δανείσει άμεσα την Ελλάδα, θα μπορούσε να δανείσει με μικρότερο επιτόκιο, αλλά φαίνεται το απαγορεύουν τα κείμενα. Πας πως τώρα είναι ώρα να ανοίξουμε τα χαρτιά και καλό θα είναι κάποια στιγμή το Κοινοβούλιο να συζητήσει και να βάλει το θέμα αυτό στο τραπέζι. Το πρόγραμμα σωτηρίας δεν λύνει βέβαια το πρόβλημα. Δεν θέλω να παρανοηθώ σε αυτά που λέω. Με ανησυχεί ιδιαίτερα αυτό που λέμε η βιωσιμότητα των δημοσίων οικονομικών και ελπίζω σήμερα το απόγευμα να καταλήξουμε σε συμβιβασμό για την έκθεση πρωτοβουλίας για την οποία είμαι αρμόδιος. Δηλαδή, το πρόγραμμα λιτότητας που επιβάλλεται σήμερα στην Ελλάδα και σε άλλους με στόχο επάνωδο σχεδόν στην δημοσιονομική ισορροπία μετά από δύο ή τρία χρόνια θα ήταν κατάλληλο θεωρητικά και το υπογραμμίζει αυτός ο οικονομολόγος αν ζούσαμε μια κατάσταση εξόδου από την κρίση δηλαδή αν ήμασταν σε κατάσταση πλήρους απασχόλησης στην περίπτωση αυτή σύμφωνα απόλυτα αν είχαμε πλήρη απασχόληση όπως γινόταν στο τέλος της δεκαετίας του 90 θα έπρεπε να δώσουμε τα πρωτογενή πλεονάσματα του προπολογισμού για τα χρέη. Και είμαι ο πρώτος που επικρίνω τη χώρα μου, τη Γαλλία, που δεν το έκανε τότε. Δηλαδή, θα έπρεπε τότε να δώσουμε το πλεόνασμα του προπολογισμού προς ε, ε, ε, ελάφρυση του χρέους. Αλλά, αγαπητοί συνάδελφοι, έχουμε βγει σήμερα από την κρίση. Στην Επιτροπή κρίση, ακούσαμε σε ακρόαση πολλούς μακροοικονομολόγους που μα εξήγησαν ότι δεν βρισκόμαστε σε κατάσταση πλήρου απασχόλησης, Είμαστε σε κατάσταση υποαπασχόλησης που σημαίνει ότι το δυναμικό παραγωγής υποαπασχολείται, υποχρησιμοποιείται, συγγνώμη. Με αυτά τα δεδομένα λοιπόν, πώς ένα πρόγραμμα λιτότητας μπορεί να αυξήσει το δυναμικό παραγωγής μιας οικονομίας Και δεν μιλάω μόνο για την Ελλάδα, μιλάω για όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Πώς ένα πρόγραμμα λιτότητας μπορεί να αυξήσει λοιπόν την δυνατότητα, του δυναμικού παραγωγής μιας χώρας, άρα να της επιτρέψει να μειώσει το χρέος. Αυτό είναι αδύνατο. Όταν μια επιχείρηση συγκεκριμένα χρησιμοποιεί 7 μηχανήματα από τα 10 που έχει, όπω συμβαίνει σήμερα, αν μειωθεί η ζήτηση, παραγγελίες, τι θα κάνει, θα επενδύσει σε ενδέκατο μηχάνημα. Όχι βέβαια, θα διαγράψει το δέκατο μηχάνημα, θα μειώσει το δυναμικό παραγωγής της. Και αυτό ακριβώς θα γίνει. Και γίνεται ήδη στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες. Κατά από αυτές τις συνθήκες λοιπόν, αν μειώνεται οι επενδύσεις, αν η κατανάλωση μειώνεται, είναι δύσκολο να υπάρξουν πρωτογενή πλεονάσματα στον προπολογισμό και να κάνω εξαίρεση για την Ελλάδα και να δω την Ισπανία. Να πάρουμε την Πορτογαλία που ήταν καλοί μαθητέ. Η Ισπανία ήταν ο πιο καλό μαθητή όσον αφορά τη δημοσιονομική πειθαρχία. Σήμερα, αν εφαρμόσετε πρόγραμμα λιτότητα στην Ισπανία, θα καταλήξετε ακριβώ το αντίθετο. Τι να μιλήσω πιο γρήγορα, τι μου λέτε, Πρόεδρε, τι μου λέτε. Να, να, να κλείνετε, διότι ο Επίτροπο θα έρθει σε 11 ώρα. Ωραία, επιταχύνω λοιπόν. Θα πετύχετε το αντίθετο αποτέλεσμα θα αυξηθεί το έλλειμμα. Και ένα τελευταίο σημείο, τα εξωτερικές ανισομέρειες που αρέσει το θέμα αυτό στο Γκίγκολτ. Σήμερα το μειοφύσιμο πρόγραμμα λιτότητας δεν λύνει τα εξωτερικές ανισοζύγιο της Ευρωζώνης. Δεν έχω χρόνο βέβαια. Όταν έχουμε ε, αρνητικό τέτοιο, μη ισορροπία, υπάρχουν τρει τρόποι. Μία είναι υποτίμηση. Δεν το θέλουμε γιατί έχουμε το ίδιο Δεν το θέλουμε. Δεύτερο τρόπο να βγει κανεί από αυτό το πρόβλημα είναι να δοθούν πόροι του προπολογισμού για να ρυθμιστούν τα σύμμετρα σοκ. Το σύμφωνο σταθερότητα σήμερα βαρύνει του εθνικού προπολογισμού. Άρα μένει μία λύση από τι τρει που είναι η χειρότερη, που είναι η μείωση των μισθών. Και αυτό κάνουμε σε όλε τι χώρε αυτή τη στιγμή. Είναι η χειρότερη λύση διότι οδηγεί σε μείωση της ζήτησης Πρόεδρο, συγγνώμη, συγγνώμη, συγγνώμη πρέπει να τελειώνετε. Τελειώνω με την εξή φράση. Ναι, καλή είναι η βιωσιμότητα των δημοσίων οικονομικών, αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση πρέπει να είμαστε ρεαλιστέ, διότι η υπερβολική τότε θα οδηγήσει στο αντίθετο αποτέλεσμα. Πρόεδρο. Συγγνώμη, αλλά χρησιμοποίησατε πέντε λεπτά. 8 λεπτά είχαμε, αλλά και όλα πήρατε πέντε λεπτά. Εξηγήστε τώρα στους άλλους γιατί δεν θα έχουν χρόνο να μιλήσουμε. Ζαν Πολ Γκοζές. Δυστυχώς θα χρειαστεί να ξαναμιλήσουμε για τα θέματα αυτά. Για να δώσω λοιπόν στον Μάρκους λίγο χρόνο, εγώ λέω θα μιλήσω σε κάποια άλλη χρονική στιγμή. Δυστυχώς όπως λέω θα έχουμε την ευκαιρία να επανέλθουμε σε όλα αυτά. Ευχαριστώ Ζαν Πολ. Ο Μάρκος πάρα πολύ σύντομα. Ευχαριστώ πάρα πολύ σύντομα κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι όλοι έχουμε καταλάβει τι σημαίνει αυτό το οποίο είχαμε συμφωνήσει πριν από 12 χρόνια. Το ευρώ και το σύμφωνο σταθερότητος δεν μας βοηθούν να λύσουμε αυτό το πρόβλημα. Τι θα είχαμε πετύχει εάν είχαμε αφήσει το ευρώ να χάσει την αξία του. Δεν νομίζω θα είχαμε λύσει το τωρινό πρόβλημα. Μια τελευταία παρατήρηση την οποία θα ήθελα να κάνω εγώ. Εγώ ήδη εξεγείρομαι για αυτά που λένε οι συνάδελφοί μου από τη Γερμανία οι οποίοι λένε ότι απέτυχε το σύμφωνο σταθερότητας. Ήδη είχαν ζητήσει πολύ από το 2004 να μειωθεί η αυστηρότητα του Συμφώνου Σταθερότητα για να μην τιμωρηθεί η Γερμανία, η οποία έχει ήδη ξεπεράσει τα όρια του. Λοιπόν, αυτά τα λίγα ήθελα να πω. Ευχαριστώ πολύ. Η Ευχαριστώ πάρα πολύ σύντομα. Πρώτα απ' όλα ήθελα να επισημάνω ότι δεν υπάρχει καμία αμφιβολία στη Σόφη ότι η βασική αιτία για το πρόβλημα που αντιμετωπίζει σήμερα η Ελλάδα είναι η ελληνική και η σημερινή κυβέρνηση κάτι κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να εξηγήσει ακριβώς τους Έλληνες πολίτες ότι η βασική ευθύνη είναι λάθη, ολιγορίες και παραλήψεις δεκαετιών που οδήγησαν στη σημερινή ε, κατάσταση. Άλλωστε αυτό είναι ο μοναδικός τρόπος για να κινητοποιήσεις τους πολίτες και να τους βάλεις αυτή τη διαδικασία της πολύ δύσκολης περίοδου που έχουμε μπροστά μας. Όμως, από την άλλη πλευρά, εάν δεν σταματήσουν επιθέσεις και σχόλια σχεδόν ρατσιστικού τύπου εναντίον των Ελλήνων και του ελληνικού λαού συλλήβδην. Ότι είναι κλέφτες, απατεώνες, τεμπέληδες. Αυτά είναι που γεννούν αισθήματα απογοήτευσης απέναντι στους Έλληνες πολίτες και βεβαίως είναι εντελώς αντιπαραγωγικά σε ό,τι αφορά την διαδικασία πειθούς αυτών των ανθρώπων να μπουν σε αυτήν την δύσκολη περίοδο που έχουμε μπροστά μας ε, με δεδομένο ότι θα έχουμε στο βάθος του τούνελ θα υπάρχει μία προοπτική. Και έρχομαι και με αυτό ολοκληρώνω κυρία Πρόεδρε ε, και στο σχόλιο που έκανε πριν ο Ζωζέ Μανουέλ, αυτός ο μηχανισμός στήριξης που συμφωνήθηκε την Κυριακή και αναμένεται να επικυρωθεί και από την Σύνοδο Κορυφής, έχει ως βασικό στόχο να δώσει στην Ελλάδα μία ανάσα που λέμε από τις επιθέσεις των αγορών, δηλαδή ε, να της δώσει την χρονική δυνατότητα για ένα διάστημα να εφαρμόσει αυτό το πολύ σκληρό πρόγραμμα που συμφωνήθηκε με στόχο, όπως είπε χθε όχι εγώ, ο Αντιπρόεδρος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου να επιστρέψει η Ελλάδα στις αγορές το ταχύτερο δυνατόν. Μπορεί να μην χρειαστεί καν να εκταμιευθεί το σύνολο των ποσών που έχουν δεσμευθεί στο πλαίσιο του μηχανισμού στήριξης. Όμως, αγαπητοί συνάδελφοι, για να συμβεί αυτό το οποίο επιθυμούμε όλοι και πρωτίστως η Ελλάδα, θα πρέπει να συνυπολογίζουμε στις παρεμβάσεις μας και τις τοποθετήσεις μας ορισμένα πράγματα. Κυρίως να μην αναιρούμε εμείς, όπως έγινε το προηγούμενο τρίμηνο, το βασικό στόχο αυτού του μηχανισμού. Με αυτή την έννοια ασφαλώς ο καθένας έχει τη δυνατότητα να ασκήσει να παρακολουθεί και θα παρακολουθούμε όλη την πορεία εφαρμογής. Αλλά δύο 24 ώρα μετά τη συμφωνία να λέμε ότι τα μέτρα δεν θα είναι αρκετά, ότι θα χρειαστεί η Ελλάδα να προχωρήσει σε διάρθρωση του χρέους της, με ορίζοντας στο τέλος την έξοδο από τη ζώνη του ευρώ, αυτού του είδους τα σχόλια ούτε τα μέτρα πρόκειται να επιτρέψουν ποτέ να εφαρμοστούν, ούτε τους Έλληνες πολίτες κινητοποιούν για να μπουν σε αυτή την ε, πολύ δύσκολη διαδικασία και εν τέλει θα μου επιτρέψετε να πω με βάση και αυτά που παρατηρούμε τις τελευταίες μέρες ουδόλως είναι προς το συμφέρον της Ευρωζώνης και της σταθερότητας του ευρώ συνολικά. Και ένα τελευταίο σβέν που συνδέεται με αυτό που σας είπα τώρα, εάν είχαμε δείξει από τις 11 Φεβρουαρίου την αποφασιστικότητα και τη στεναρότητα που μπορούσαμε και έπρεπε να δείξουμε, πιστεύω, αυτή είναι η πεποίθησή μου, μπορεί να κάνω λάθος, ότι αυτός ο μηχανισμός στήριξης θα μπορούσε όντως να λειτουργήσει αποτρεπτικά. Δηλαδή να μην χρειαστεί να εκταμιευτούν τα κονδύλια που εκταμιεύονται τώρα. Η Ελλάδα το Φεβρουάριο δανειζόταν με 6% επιτόκιο, 1% λιγότερο από αυτό που προβλέπεται από το μηχανισμό στήριξης και στη διάρκεια των τελευταίων εβδομάδων τα επιτόκια φτάσανε στο 10%. Δεν επιδεινώθηκε η κατάσταση της ελληνικής οικονομίας μέσα σε λίγες εβδομάδες με τρόπο που να δικαιολογεί αυτή τη διαφορά στα επιτόκια. Ευχαριστώ πολύ. Thank you very much, Annie. Thank you, colleague. Ευχαριστώ, Άννη και αγαπητοί συνάδελφοι. Εν πολύ συντομία, στο τέλος της συζήτησής μας, ήθελα να πω ότι καταδεικνύει αυτή η συζήτηση ότι τα μέλη του Κοινοβουλίου και της Επιτροπής μας γνωρίζουν ποια είναι τα προβλήματα, ποιε είναι οι ευαισθησίες και είναι απόλυτα ικανοί να είναι μια φωνή αλληλεγγύης και σοφροσύνη σε σχέση με την επίλυση των προβλημάτων της Ελλάδος. Σας ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ συνάδελφοι και πάω τώρα να βρω τον κύριο Επίτροπο. Um, λοιπόν, <clears throat> νιώθω μεγάλη χαρά. Παρακαλώ οι ιδιωτικέ συζητήσει μπορούν να, συζητήσουν, να σταματήσουν. Ευχαριστώ πολύ. Χαίρομαι πάρα πολύ μπορώ μπορούμε να υποδεχθούμε τον Επίτροπο κ. Μπαρνιέ στην Επιτροπή μας. Τον καλωσορίζω θα έπρεπε να έχει γίνει αυτή η συνάντηση το Στρασβούργο, αλλά ορισμένοι από εμά ήμασταν ηφαιστειόπληκτοι. Είναι η πρώτη φορά λοιπόν που είχαμε τη δυνατότητα να χαιρετήσουμε τον κύριο Επίτροπο στην Επιτροπή μας. Προφανώς είχε έρθει όταν είχαμε τη συνάντηση με τα Εθνικά Κοινοβούλια, αλλά αυτή είναι η πρώτη φορά που έρχεται αμυγός ενώπιον της Επιτροπής μας για να μας ενημερώσει για τα τελευταία στοιχεία εξελίξεων στις χρηματαγορές και να απαντήσει στα ερωτήματά μας. Πολύ χαιρόμαστε που σας έχουμε εδώ κύριε Μπαρνιέ. Ξέρουμε ότι είναι η πρώτη φορά, αλλά θα ακολουθήσουν και άλλες. Και έχετε το λόγο κύριε Επίτροπε. Κυρίε και κύριοι βουλευτές, καλημέρα σε όλους σας. Για πολλούς λόγους χαίρομαι πάρα πολύ που με ενωπιών σας. Θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Πρόεδρο για την ε, υποδοχή που με επιφυλάξετε. Κυρίε και κύριοι, χωρίς να καταδαπανίσω το χρόνο σας. Θέλω να είμαι στον τον πιο εξαντλητικό στην αρχική μου παρέμβαση προτού απαντήσω στα ερωτήματά σας. Μετά από τη μεγάλη αναταραχή του 2008 ελήφθησαν πολλές αποφάσεις, ξεκίνησαν πολλές προσπάθειες αναζήτησης νέων λύσεων. Αρκεί να δει κανείς τις εφημερίδες, τις χθεσινές, τις σημερινές, βλέπουμε ότι η κρίση των αγορών εξακολουθεί να υπάρχει. Διατηρείται αυτή η κρίση ε, αφορά τις επιχειρήσεις, αφορά τους ηγέτες των επιχειρήσεων, τους πολιτικούς, τους πολίτες που πολλές φορές έχουν κάθε λόγο να είναι ανήσυχοι, απέχουμε πόρο από το να έχουμε εξέλθει από την κρίση. Είχα πει τον Ιανουάριο ότι η πεποίθησή μου είναι ότι δεν πρόκειται να βγούμε από την κρίση αυτή στην ίδια κατάσταση στην οποία είχαμε μπει, ούτε σε ό,τι αφορά τη ρύθμιση των αγορών, και θα επανέλθω, ούτε σε ό,τι αφορά την ε, ανάπτυξη την οικονομική, την φύση και την ποιότητα αυτής της οικονομικής ανάπτυξης πρέπει να είναι πιο ισορροπημένη, πιο ισοδίκαια και που να σέβεται ιδιαίτερα και το περιβάλλον. Αλλά δεν είναι ακριβώς η κατάλληλη στιγμή να σταθούμε μονάχα στα λόγια και να μείνουμε άπρα χωρίς, ε, χωρίς κάποια δράση. Θα πρέπει να αποφασιστούν οι συνέχειες που θα δοθούν θα πρέπει η Ευρώπη να καταλάβει τα διδάγματα της κρίσης και θα πρέπει να ακολουθήσουμε ένα συγκεκριμένο δρόμο. Είχα ζητήσει από, από τον Ιανουάριο ήδη το έργο της ε, εποπτείας, το εγχείρημα της εποπτείας να γίνει με έναν τρόπο ευφυή με τη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είχαμε και πολλές ευκαιρίες να <clears throat> ανταλλάξουμε απόψη για τα θέματα αυτά. Θέλω λοιπόν εκ βάθους καρδίας να σας ευχαριστήσω για τη συμμετοχή σας. Είναι φορτωμένο το νομοθετικό χρονοδιάγραμμα και μέσα στον επόμενο χρόνο, μέχρι την επόμενη άνοιξη δηλαδή, του 2011, θα πρέπει να εκπληρώσουμε όλες αυτές τις υποχρεώσεις που ανέλαβαν οι G20 και να υπάρξουν ε, στα χέρια του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου προτάσει νομοθετικέ που υλοποιούν τι δεσμεύσει που ανέλαβαν οι ηγέτε τη Ευρωπαϊκή Ένωση στην συνεδρία των G20. Γιατί πρέπει να δράσουμε τώρα. Το λέω ότι είναι κομβική οι επόμενοι μήνες για την επιβίωση του χρηματοοικονομικού μας συστήματος και εξάλλου είναι κομβική για το σύνολο της οικονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θέλω να χαιρετήσω το ιδιαίτερα σημαντικό έργο της Επιτροπής ΚΡΙΣ με επικεφαλής τον Wolfgang Κρίς και την έκθεση της κυρίας Περβάνος Μπερές. Το 2010 θα πρέπει να είναι το έτος <clears throat> που θα υπάρξει η απαρχή της οικονομικής ανάκαμψης, το ελπίζουμε, θέλουμε να είμαστε προσεκτικοί και επιφυλακτικοί, ακόμα και αν υπάρχουν θετικά στοιχεία, αυξάνει πιο γρήγορα η βιομηχανική παραγωγή και μπορούμε να φτάσουμε ένα επίπεδο 4% στην οικονομική ανάπτυξη. Μπορεί να επανέλθει λοιπόν η εμπιστοσύνη στις ε, επιχειρήσεις και μπορούμε ιδιαίτερα να δούμε ότι υπάρχουν θετικά στοιχεία για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και την χρηματοδότησή τους. Αλλά μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι δεν θα επανέλθει η κρίση, ότι θα επανέλθουμε στο επίπεδο παραγωγής πριν από την κρίση. Έχουμε ανισορροπίες στην παγκόσμια παραγωγή που έχουν οξυνθεί. Το 2010 ήταν επίσης κυρίες και κύριοι το έτος που έγινε σαφές ο αντίκτυπος της κρίσης στον προϋπολογισμό των κρατών μελών <clears throat> που θα πρέπει τώρα να αντιμετωπίσουν τεράστια προβλήματα που απαιτούν άμεσες παρεμβάσεις. Πρέπει να υπάρξει μια άμεση παρέμβαση λοιπόν σε όλους τους τομείς για να αντιμετωπιστεί το σοκ της ε, έλλειψης ανάπτυξης και η άνοδος της ανεργίας. Όλοι οι πολίτες, όλοι οι φορολογούμενοι έχουν με κάποιο τρόπο πληγή από τα, από τα συνέπειες των σφαλμάτων που διέπραξαν ορισμένε τράπεζες στο χρηματοπιστωτικό τομέα και το γεγονός ότι έχουν χάσει και τον μπούσουλα οι <clears throat> επικεφαλής <clears throat> των ε, κρατών μελών και κυβερνήσεών μας. Πιστεύω λοιπόν ότι βλέπουμε αυτή τη στιγμή να υπάρχει ανησυχία των αγορών για την κατάσταση των δημοσίων οικονομικών στην Ευρώπη και σε άλλα μέρη του κόσμου. Πολλές φορές αυτή η ανησυχία οδηγεί σε σοβαρά προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν με μια κοινή δράση ανηλεγγύης όπως αυτή που έχουμε οικοδομήσει έναντι ενός από τα κράτη-μέλη μας, έναντι της Ελλάδος. Δεν θα επανέλθω τώρα λεπτομεριακά στα θέματα της Ελλάδος που είναι περισσότερο στην αρμοδιότητα του συναδελφού του κ. Όλιρεν. Πρέπει όμως να αντλήσουμε κάποια συμπεράσματα σε ό,τι αφορά τις αγορές και τους χρηματοοικονομικούς εμπλεκόμενους, τους φορείς πιστοληπτικής ικανότητος. Πρέπει εδώ να εξασφαλίσουμε και την υπευθυνότητα και την διαφάνειά τους. Είναι λογικό οι φορείς αυτοί να αξιολογούν την κατάσταση των κρατών, αλλά θα πρέπει να ξέρουν και ποιες είναι οι συνέπειες των αποφάσεων που παίρνουν και αυτό θα πρέπει να σημαίνει ότι θα πρέπει να έχουν μια υπευθυνότητα και να λειτουργούν με έναν τρόπο ιδιαίτερα διάφανο. Γι' αυτό εμείς θέλουμε να εξασφαλίσουμε και μεγαλύτερο ανταγωνισμό και πολυμορφία στον τομέα των φορέων πιστοληπτικής αξιολόγησης. Η εφαρμογή λοιπόν των ρυθμίσεων που έχουμε εγκρίνει για τον τομέα αυτό, που θα αρχίσουν να λειτουργούν από το Δεκέμβριο του 2010, θα μας επιτρέψουν να προχωρήσουμε προς την κατεύθυνση μεγαλύτερης διαφάνειας και μεγαλύτερης υπευθυνότητας. Αλλά αρκεί αυτό. Δεν ξέρω, αλλά πολύ γρήγορα θα προβούμε σε μια αξιολόγηση της, των επιπτώσεων αυτής της οδηγίας για τους οίκους πιστοληπτικής αξιολόγησης, για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε και περαιτέρω. Στον χρηματοοικονομικό τομέα, το 2010 διαγράφεται σαν έτος επαν, επανόδου της κερδοφορίας. Αυτό είναι θετικό, αλλά μόνο αν αυτό αφορά όλες τις οικονομίες που χρειάζονται χρηματοδότηση. Ελπίζω ότι αυτό δεν θα οδηγήσει και πάλι σε αλόγιστη προσφυγή σε ανάληψη κινδύνων, όπως είδαμε στο παρελθόν. Πρέπει τα μπόνους των στελεχών να υπόκειται σε αυστηρούς κανόνες στο μέλλον. Και όλα αυτά με οδηγούν στο κύριο μήνυμα το οποίο θέλω να σας δώσω, το 2010 θα πρέπει να είναι και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα είναι το έτος που θα εφαρμόσουμε όλες τις δεσμεύσεις που έχουμε αναλάβει στο G20 για να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε μεγαλύτερη χρηματοοικονομική ισορροπία. Οι Αμερικανοί παρτενέρ εργάζονται και αυτοί σε, για να πετύχουν τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις για τη ρύθμιση και την εποπτεία των αγορών και φαίνεται να έχουμε καλούς ιονούς ότι θα μπορέσει να υπάρξει και μια συμφωνία για μια μεταρρύθμιση άξια του ονόματός της. Όλη την επόμενη εβδομάδα θα, θα είμαι στι Ηνωμένε Πολιτείε. Για 4,5 μέρες συναντήσεων και είμαι πεπισμένο ότι ο διεθνή συντονισμό μπορεί να ενισχύσει τις μεταρρυθμίσεις μας και δεν θα πρέπει να είναι ένα πρόσχημα για να τις αποδυναμώσουμε τις μεταρρυθμίσεις ή να τις αναβάλουμε. Και θα συνεχίσω τις προσπάθειες αυτές και την επόμενη εβδομάδα με τους Αμερικανούς ομολόγους μας, γιατί μόνο από κοινού μπορούμε να αντλήσουμε συμπεράσματα για την κρίση και μόνο έτσι μπορούμε να καταλήξουμε σε σωστές λύσεις και όχι σε κατακαιρματισμένες ή αντιμαχόμενες λύσεις. Εμείς δεν έχουμε το δικαίωμα να υποβάλουμε τους πολίτες και τους φορολογούμενους σε πρόσθετα βάρη και κυρίως δεν πρέπει να χάσουμε το ραντεβού του 2010, του οποίου τόνισα τη σημασία. Και έχουμε τώρα στις προτάσεις για τις οποίες πρέπει να συνεργαστούμε. Έχουμε είναι απαραίτητο να έχουμε τα μέσα για τη δράση αυτή με την συνθήκη της Λισαβόνας, με τη δυνατότητα των θεσμικών οργάνων να λειτουργήσουν προς την κατεύθυνση αυτή, ιδίως την Κομισιόν και το Κοινοβούλιο. Ό,τι και να λένε ορισμένοι, η Ευρωπαϊκή Ένωση έδειξε και πάλι αυτό το Σαββατοκύριακο ότι μπορούσε να βρει λύσεις ενώπιον κρίσεων πρωτοφανών και ότι η Ευρωπαϊκή Αλληλεγγύη υπάρχει. Αλλά τα γεγονότα αυτά μας τονίζουν επίσης και την ανάγκη του να τηρήσουμε τις υποχρεώσεις μας να μην ξεχάσουμε τα διδάγματα της κρίσης, να μην αφήσουμε να αυξάνονται οι αποκλίσεις απόψεων μεταξύ μας ή μεταξύ θεσμικών οργάνων, μεταξύ κρατών, γιατί όλοι έχουμε τις ίδιες ευθύνες. Σας προτείνω λοιπόν να εργαστούμε το επερχόμενο έτος σε μία σειρά από προβλήματα. Το κυριότερο από αυτά είναι το θέμα μιας καλύτερης εποπτείας, μιας πιο ευρωπαϊκής εποπτείας του χρηματοπιστωτικού τομέα. Αυτό αποτελεί ένα από τα θεμέλια της κοινή μας προσπάθειας για να εξασφαλίσουμε τη ρύθμιση των αγορών και θέλω να συνεργαστώ μαζί σας για να μπορέσουμε να τηρήσουμε τα δύσκολα αλλά απαραίτητα χρονοδιαγράμματα της 1 η Ιανουαρίου 2011 ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει ένα σύστημα εποπτείας άξιο του ονόματός του ξεκινώντας από μια κοινή προσέγγιση του Συμβουλίου που υπάρχει ήδη στο Κοινοβούλιο το σύνολο των εισηγητών Σκίνερ, Γκουλάρ, Μαργάγιο, ε, Πρεσέδο έχουν προσθέσει σημαντικές ιδέες σε αυτή τη συζήτηση που θα συνεχίσει βέβαια και τις επόμενες μέρες και με την ευκαιρία της ψηφοφορία που θα κάνετε ως ονούπο πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορέσει να διατηρηθεί μια συνεκτικότητα στην προσέγγιση και στο επίπεδο φιλοδοξίας. Βλέπω τη δική σας θέση που είναι πολύ κοντά με τη θέση της Κομισιόν και τη θέση του Συμβουλίου που βέβαια είναι διαφορετικές μεταξύ τους. Υπάρχουν αποκλήσεις αλλά υπάρχουν και δυνατότητες συμφιλίωσης αυτών των αποκλεινουσών απόψεων και είναι ρόλος της Κομισιόν και δικός μου να εργαστούμε για την σύγκληση μεταξύ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου αν υπάρξει και από τις δύο πλευρές πνεύμα ανοιχτό και πνεύμα ευκαμψίας. Όλα αυτά θα μας οδηγήσουν σε μια προσθέμενη αξία, σε ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τον χρηματοπιστωτικό τομέα στην Ευρώπη, να είμαστε η πρώτη περιοχή του κόσμου που έχει ένα τέτοιο μοντέλο ρύθμισης και εποπτείας. Δεύτερη προτεραιότητα, η ρύθμιση των χρηματαγορών και των εμπλεκόμενων στις αγορές. Κανείς δεν πρέπει να ξεφύγει από αυτήν την εποπτεία και τη ρύθμιση. Έχουμε δύο πράγματα που πρέπει να κάνουμε το 2010, να βρούμε μια συμφωνία για την απαραίτητη ρύθμιση ε, φορέων όπως είναι τα κεφάλαια ε, equity, τα ιδιωτικά κεφάλαια και οι, τα hedge funds. Εκεί πέρα υπήρξαν σημαντικές πρόοδοι οι ε, οποίες επετέφθησαν και χαιρετίζω το έργο του Ζαν Πιερ Γκοζές. Χρειάζεται και μια συμφωνία μεταξύ των θεσμικών οργάνων το ταχύτερο δυνατό ή δυνατόν πριν από το καλοκαίρι. Για τις τρίτες χώρες επίσης, που αυτό παραμένει από τα δύσκολα θέματα, θα ήθελα να μειωθεί η ανάγκη να υπάρξει ισότητα των διαχειριστών κεφαλαίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση έναντι αυτών των τρίτων χωρών, θα πρέπει να υπάρχουν ίσες προδιαγραφές και ίσες προϋποθέσεις. Και εμείς θα εξετάσουμε νέες προτάσεις για να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε ένα αποτελεσματικό σύστημα εξίσωσης. Και επέκεινα αυτών των κειμένων χρειάζεται να υπάρξει και ένα νομοθέτημα το οποίο να ρυθμίζει τα παράγωγα προϊόντα στις χρηματαγορές που είναι απαραίτητο για τη σταθερότητα των αγορών. Εγώ θα προτείνω μια στρατηγική πρωτοβουλία για τα παράγωγα η οποία αφορά και τα ποσά τα οποία διακυβεύονται και τα προϊόντα τα οποία κυκλοφορούν στις αγορές θα είναι στρατηγικού χαρακτήρα γιατί κάθε μήνα σχεδόν βλέπουμε να αναδύονται νέα παραδείγματα σε πολλούς τομείς που μας αναγκάζουν να σκεφτούμε για το αν λειτουργούν σωστά αυτές οι αγορές. Όλα αυτά κάνουν ισχυρότερη την αποφασιστικότητά μου να σας προτείνω μια πιο αποτελεσματική ρύθμιση για τα κρατικά ομόλογα κάνουμε μία μελέτη της αγοράς αυτής κρατικών ομολόγων παρακολουθώντας τις κινήσεις των τελευταίων μηνών. Δεν θέλω να αποκαταλάβω τα συμπεράσματα, αλλά νομίζω ότι πρέπει να εξασφαλίσουμε τη διαφάνεια, την απόλυτη διαφάνεια αυτών των αγορών, ώστε να μπορούν και οι ρυθμιστές να εξασφαλίζουν την καλή τους λειτουργία και να δρουν σε περίπτωση που υπάρχουν ελλείψεις και προβλήματα. Πριν από το τέλος του έτους θα πρέπει να έχουμε αυτό το γενικό κείμενο σε σχέση με τα παράγωγα προϊόντα για την τυποποίηση και, την, ε, τον κεντρικό συμψηφισμό αυτών των προϊόντων κάτω από αυστηρή εποπτεία. Πρέπει λοιπόν να υπάρχει και καταγραφή των συναλλαγών παραγόγων σε κεντρικά μητρώα συναλλαγών για να υπάρξει και καλύτερος, καλύτερη παρακολούθηση για τα θέματα αυτά. Ξέρω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει πάρει ένα πρωτοπόρο ρόλο χάρη στην έκθεση του Βέρνερ Λάγκεν και χάρη στις τροπολογίες που καταθέσατε πολλοί από εσά και χάρη στην ακρόαση της προηγούμενης εβδομάδας. Πιστεύω ότι οι προτάσεις μας θα λάβουν υπόψη και την ανάλυση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τα ερωτήματα τα οποία έχετε γύρει και ιδίω σε ό,τι αφορά του κανόνε, οι οποίοι προβλέπουν ότι για τις μη χρηματοπιστωτικέ εταιρείε θα πρέπει να υπάρξει διαφορετική αντιμετώπιση. Μαζί με τι υπηρεσίε μου έχω ακούσει ε, την άποψη αυτών των επιχειρήσεων, των βιομηχανικών επιχειρήσεων για τα θέματα αυτά και επίσης πρέπει να εξετάσουμε και το δυνητικό αντίκτυπο της νομοθεσίας που θα θεσπίσουμε. Είναι σαφές λοιπόν ότι πρέπει να μην υπόκειται στην ανάγκη συμψηφισμού, στην υποχρέωση συμψηφισμού, οι μη χρηματοπιστωτικέ εταιρείε. Αλλά, σαν αντιστάθμισμα, θα του ζητήσουμε να διαχειρίζονται τους κινδύνους που αφορούν τα μη συμψηφισμένα κεντρικά ε, παράγωγα και την αντιμετώπιση του συστημικού κινδύνου που προκύπτει από κάτι τέτοιο. Θα είμαστε λοιπόν επάγρυπνοι ώστε αυτή η απόφαση να μην την χρησιμοποιήσουν για να την εκμεταλλευτούν οι μη χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί και να μην προχωρήσουμε σε κάτι που θα ευνοήσει το ρυθμιστικό αρμπιτράζ. Θα πρέπει να είμαστε απόλυτα συνεκτικοί και σύμμορφοι με αυτά τα οποία γίνονται και στι ΗΠΑ. Ένα τέταρτο σημείο των μελλοντικών προτάσεων που επίκυνται είναι το λεγόμενο short selling, οι γυμνές πωλήσει ε, ε, αξιογραφών. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρξει και εδώ μια πρόταση σε σχέση με τις λεγόμενες γυμνές πωλήσει αξιογράφων που θα δοθεί στην, στην ε, δημοσιότητα τον Οκτώβριο. Δηλαδή να διατηρηθούν οι πρακτικές οι οποίες είναι χρήσιμες για τις αγορές και τους επενδυτές για να υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το μοντέλο του ΣΕΖΑ, τη Επιτροπή Ρεθνιστών, αλλά θα πρέπει να προχωρήσουμε ακόμα περισσότερο. Θα πρέπει να αποφύγουμε τα κράτη-μέλη να παίρνουν κατακαιρματισμένα εθνικά μέτρα, όπως φάνηκε να γίνεται κατά τη διάρκεια της κρίσης. Θα πρέπει να είμαστε σε θέση να επιβάλλουμε κυρώσεις στις παραβιάσεις των κανόνων. Δεν μπορεί να υπάρξει αποτελεσματικό πλαίσιο υποπτίας παρά μόνο αν όλοι οι ρυθμιστές και όλα τα κράτη-μέλη δώσουν τα απαραίτητα, την απαραίτητη υποστήριξη σε μέτρα κυρώσεως των παραβιάσεων και εδώ θα υπάρξει μια μεταρρύθμιση της οδηγίας για την κατάχρηση αγοράς που θα σας προτείνει η Κομισιόν το 2010 για να μπορέσει να καλύψει τα τωρινά κενά των οδηγιών οι οποίες ισχύουν ιδίως σε ό,τι αφορά τη χρήση πολυμερών συστημάτων ε, διαπραγμάτευσης και επίσης για ορισμένα παράγωγα τα εξωχρηματιστριακά, τα over the counter δηλαδή, securities. Ο στόχο είναι να μπορέσουν οι αρχέ μα να έχουν τα απαραίτητα μέτρα και να μπορούν να παρεμβαίνουν αν θεωρούν ότι διακυβεύεται η σταθερότητα τη αγορά και η οδηγία MIFID θα βοηθήσει την πρόοδο προ την κατεύθυνση αυτή και θα ήθελα να ακούσω και τι δικέ σα απόψει, ιδίω τη Kate Swin Brown, για τα ζητήματα αυτά. Ένα τρίτο μεγάλο θέμα που μα απασχολεί είναι το να γίνουν στερεότερε οι τράπεζε πρέπει να αντέχουν περισσότερο οι τράπεζές μας να μην υπάρξει υπερβολική ανάληψη κινδύνου από τις τράπεζες και ιδίω να τεθεί σε εφαρμογή η οδηγία κεφαλαιοχικής επάρκειας 3, σε 3, μετά το έργο της ε, Αρλέν Μακάρτιν για αυτό το θέμα που αφορά τα ίδια κεφάλαια και τις κεφαλαιοχικές απαιτήσει των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Είναι σαφές ότι σε περίπτωση Πολύπλοκη τυπλοποίηση για οι κεφαλουχικές επάρκειε που προβλεπόταν δεν ήταν επαρκή. Πρέπει να ενισχυθούν αυτοί οι κανόνε. είναι λοιπόν σημαντικέ ρυθμίσει για να γίνουν οι τράπεζέ μα στερεότερε, να παίξουν σημαντικότερο ρόλο στη διεθνή αγορά. Θα πρέπει φυσικά να εξασφαλίσουμε και την ισότητα ανταγωνισμού με του διεθνεί εταίρου μα. Αυτό είναι ένα θέμα για το οποίο θέλω να μιλήσω και με του Αμερικανού Γιατί πολλοί ανησυχούν για τις αποκλήσεις μεταξύ της εφαρμογή αυτών των μέτρων στην Ευρώπη και στις Ηνωμένε Πολιτείε. Είναι πιθανό οι νέοι κανόνες της Βασιλείας, Βασιλείας 3, θα τροποποιηθούν εν ώψη της μελέτης αντικτύπου η οποία έχει γίνει για τα θέματα αυτά. Σημερίζομαι λοιπόν τις ανησυχίες σας και μαζί με την κυρία Μακάτι και άλλους θα προσπαθήσουμε να βρούμε μια ισορροπημένη λύση. Επίσης πρέπει να αντλήσουμε και τα συμπεράσματα σε ό,τι αφορά τους κανόνες προληπτικής εποπτείας η Κομισιόν συμμετέχει στις εργασίες της Επιτροπής της Βασιλείας για να μπορέσουμε να οικοδομήσουμε ένα πιο ανθεκτικό πλαίσιο για την προληπτική εποπτεία. Και αυτό είναι μια απόφαση των G20 για να μπορέσουμε να ενισχύσουμε την ανθεκτικότητα του διεθνούς συστήματος στα χρηματοοικονομικά και να εξασφαλίσουμε ή σε συνθήκε ανταγωνισμού. Αυτά είναι τα στοιχεία της Βασιλείας 3. Όλα αυτά λοιπόν θα αποτελέσουν αντικείμενο προτάσεων στην Οδηγία Κεφαλουχικής Επάρκειας 4, σε 4, με συγητή τον κύριο Καρά. Χρειάζεται λοιπόν να γίνει και μια ευρεία διαβούλευση για τα θέματα αυτά για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τον αντίκτυπο των δυνητικών αλλαγών και να κάνουμε την σωστή τοποθέτηση, μια τριπλή λοιπόν προσαρμογή στο χρόνο σε σχέση με την χρονική στιγμή εφαρμογή τους, σε σχέση με το σωρευτικό αποτέλεσμα της εφαρμογής αυτών των μέτρων και τρίτον σε σχέση με αυτό που κάνουμε στην Ευρώπη και αυτό που κάνουν οι εταίροι μας στις ΗΠΑ. Δηλαδή οι εξωτερικές σχέσεις. Δεν πρέπει να αυτοσχεδιάσουμε, δεν πρέπει να βιαστούμε, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε όλα αυτά τα διδάγματα της καλύτερης ρύθμισης, better regulation. Η Κομισιόν θα λάβει υπόψη όλα τα στοιχεία αυτά σε ό,τι αφορά τη μικροπροληπτική και μακροπροληπτική εποπτεία. Γι' αυτό εγώ αποδίδω μεγάλη σημασία στην πλήρη αυτή διενέργεια διαλόγου πλήρους και ανοιχτού. Τέταρτη προτεραιότητα που είναι πολύ σημαντική είναι το να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε και ένα πλαίσιο διαχείρισης και πρόληψης των μελλοντικών κρίσεων στην Ευρώπη. Για να μειώσουμε τον αντίκτυπό τους και να αποφύγουμε οι πολίτες και οι φορολογούμενοι να είναι στην πρώτη γραμμή πυρός και να πληρώνουν αυτή την ύφη. πρέπει να είναι οι μέτοχοι και οι ακάλυπτοι πιστωτές οι οποίοι θα πρέπει καταρχήν να αναλαμβάνουν το βάρος αυτών των απολειών και όχι οι φορολογούμενοι. Σε όλα τα κράτη-μέλη θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα να οργανωθούν οι χρηματοπιστωτικοί πορείς με τέτοιο τρόπο ώστε να αναδιαφρώνονται προτού γίνουν αφαιρέγκοι αυτοί οι φορείς και να διατηρηθούν τα δικαιώματα των φορολογουμένων. Αυτό σημαίνει πρέπει να έχουμε μια φορολογία η οποία θα είναι και παρεμβατική, θα επιτρέπει την μεταφορά στοιχείων ενεργητικού και που μπορεί να επιβάλλει και την καταγραφή απολειών στην περίπτωση που δεν είχαν τύχει εγγύησεων. Και χρειάζεται ιδιαίτερη ρύθμιση στις διαμεθοριακού χαρακτήρα τράπεζες. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα και εμείς υποτιμούμε την πολυπλοκότητά του. Γι' αυτό πρέπει να προχωρήσουμε βήμα-βήμα. Έχουμε κάνει διαβουλεύσεις από πέρσι και έχουμε οργανώσει ε, διασκέψει για τα θέματα αυτά και στο φως των αποτελεσμάτων αυτής της διαβούλευσης θα παρουσιάσουμε μια ανακοίνωση τον Οκτώβριο σε σχέση με την πρόληψη, την εποπτεία και τη διαχείριση των κρίσεων. Ένα πρώτο σημαντικό πλαίσιο για να προχωρήσουμε θα είναι η εναρμόνιση των συστημάτων επίλυσης αυτών των προβλημάτων σε εθνικό επίπεδο. Εμείς σκεφτόμαστε ότι ίσως θα πρέπει να υπάρξει και μια ευρωπαϊκή αρχή για να εναρμονίσουμε το δίκαιο πτώχευσης, το οποίο αυτή τη στιγμή είναι κατακαιρματισμένο σε 27 εθνικά δίκαια. Ένα σύστημα λοιπόν πρόληψης θα πρέπει να βασίζεται στην αρχή ο ρηπαίνων πληρώνει. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι οι μηχανισμοί χρηματοδότησης θα πρέπει να εξασφαλίσουν ότι αυτός ο οποίος φταίει για μια κρίση θα πληρώσει πράγματι για τα αποτελέσματα της κρίσης και γι' αυτό υποστηρίζω τη δημιουργία ενός ταμείου για την ε, αντιμετώπιση των κρίσεων. Και αυτό θα παρουσιαστεί από την Κομισιόν από τον επόμενο μήνα. Ξέρουμε ότι πολλές φορές τα πρώτα θύματα είναι οι μικροκαταθέτες και οι μικροεπενδυτές. Εμείς θέλουμε να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρξει εγγύηση των καταθέσεων, αλλά παραμένουν πολλά να πράξουμε. Σας προτείνω να υπάρξει μία σε βάθος τροποποίηση αυτής της οδηγίας στο κεφάλαιο, ώστε το Ταμείο αυτό αντιμετώπιση των κρίσεων να μπορεί ήδη να χρηματοδοτείται από συνεισφορές που βασίζονται στο επίπεδο κινδύνου, να γίνονται οι πληρωμές σε λίγες μέρες και όχι σε εβδομάδες και να είναι πλήρως πληροφορημένοι καταθέτες για την κάλυψη και τα όρια κάλυψης, κάτι το οποίο θα βοηθήσει, θα βελτιώσει την ευρωπαϊκή χρηματοοικονομική νομοθεσία, αλλά θα αυξήσει και την ε, εμπιστοσύνη των καταναλωτών και φορολογουμένων. Τέλο η διακυβέρνηση των επιχειρήσεων. Υπάρχουν ορισμένα προβλήματα τα οποία θα πρέπει να αντιμετωπιστούν στη ρίζα του. Θα πρέπει να αναφερθώ λοιπόν στι τράπεζε, στι ασφαλιστικέ εταιρείε και του άλλου παίκτε του χρηματοοικονομικού τομέα που έδρασαν με τρόπο αλόγιστο και άφρονα. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρξει μια πιο σωστή πολιτική αποδοχών των υψηλών στελεχών και όχι αυτή η οποία οδήγησε σε αγανάκτηση της κοινή γνώμης. Χαιρετίζω λοιπόν τις διατάξεις της εκθέσεως της κυρίας Μακάτη σε σχέση με την ε, αμοιβή των στελεχών σε περιπτώσεις επίσης αποχώρησης και την ε, ε, ορθή αντιμετώπιση αυτών των θεμάτων. Η πρότασή μα είναι από το Μάιο η Κομισιόν να εγκρίνει μια πράσινη βίβλο η οποία διερευνά του τρόπου με του οποίου θα ενισχύσουμε την διακυβέρνηση των επιχειρήσεων, καταρχήν στου χρηματοοικονομικού φορεί και θα δράσουμε στη συνέχεια. Αλλά σα είπα ήδη ότι θα πρόκειται για μέτρα ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών και τη διαχείριση των κινδύνων στους χρηματοοικονομικούς φορείς που αυτό θα πρέπει να είναι ευθύνη των ίδιων των επιχειρήσεων. Θέλουμε αυτοί τα στελέχη των επιχειρήσεων να έχουν την εμπειρογνωμοσύνη και τον απαραίτητο χρόνο για να εκπληρώσουν το έργο τους, δηλαδή πρέπει να είναι στελέχη ικανά. Σε δεύτερο επίπεδο, σε δεύτερο χρονικό επίπεδο, θα αντιμετωπίσουμε το θέμα της ευκυβερνησίας στις εισηγμένες στα χρηματιστήρια επιχειρήσεις και το θέμα της κοινωνικής τους ευθύνης. Αυτά λοιπόν κυρία Πρόεδρε, ευχαριστούμε για την προσοχή σας και την υπομονή σας. Νομίζω ότι με τον τρόπο αυτό έχω σεβαστεί τις ε, υποχρεώσεις μου ενώπιόν σας, εξηγώντας με τον πιο πλήρη τρόπο το χρονοδιάγραμμα των εργασιών μας και υπογραμμίζω μια ακόμα φορά το ότι αυτό το οποίο με ενδιαφέρει είναι να αντιμετωπίσουμε το χρόνο που περνάει ανάμεσα στην έκρηξη της κρίσης, κρίσης που δεν έχει ξεπεραστεί και τη λήψη των αποφάσεων, ιδίως στην υλοποίηση των αποφασίσεων του Pittsburgh των G20 και το να είναι πραγματικά λειτουργικά τα μέτρα αυτά. Μόνο σε ορισμένου τομεί έχουμε προχωρήσει. Προ το παρόν είμαστε περιορισμένοι σε ό,τι αφορά την εφαρμογή αυτών των μέτρων. Θέλω να είναι άψογη η Κομισιόν σε σχέση με αυτά που απαιτούνται από αυτήν για την εφαρμογή των αποφάσεων του G, των G20, το ταχύτερο δυνατό. Και εγώ, όπω είναι ο ρόλο μου, είμαι έτοιμο να συνεργαστώ και με το Συμβούλιο και με το Κοινοβούλιο, ώστε η εφαρμογή σε λειτουργικό επίπεδο αυτών των αποφάσεων να μην βραδιπορήσει υπερβολικά. Αυτά λοιπόν για το πνεύμα και το πλαίσιο εργασία το οποίο σα προτείνω κυρίε και κύριοι βουλευτέ, το οποίο θα είναι και αντικείμενο περαιτέρω συζητήσεων μεταξύ ημών και ημών με ύψιλον τι επόμενε μέρε. Ευχαριστώ. Uh, thank you, I, I... Ευχαριστώ τον Επιτροπό. Πραγματικά είναι Πολύ εντατικό το πρόγραμμα εργασία σα. Δεν είχαμε βέβαια καμία αμφιβολία γιατί το παρακολουθούμε στενά. Ήδη 14 μέλη έχουν εγγραφεί στον καταλογό μου, μόλι έγιναν 15. Οπότε να τα δούμε λίγο ομαδοποιημένα. Α, 16 τώρα. Ένα θέλω να σας ζητήσω εγώ. Δεν είπατε έτσι ε, παρόδο την οδηγία για το IFM Μιλήσατε όμως και για τα hedge funds και ξέρω ότι αυτό πραγματικά την χάνει μεγάλης προσοχής από τα ΜΜΕ και πολλά από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε και κάποια κράτη-μέλη δεν είναι ικανοποιημένα, είναι γιατί πραγματικά ε, ε, επεκτείνεται πέραν αυτών των επιχειρήσεων και ομήλων αυτή η, αυτό το χαρτοφυλάκιο. Οπότε θα μπορούσατε να μας πείτε κάτι παραπάνω. γιατί επηρεάζει πολύ και τα καταπιστεύματα και τα συνταξιωτικά ταμεία και πολλά άλλα ταμεία τα οποία κάποιοι θεωρούν αθώα στα, ενώ μέσα στην όλη αυτή, στον όλο κυκαιώνα της οικονομικής κρίσης. Λοιπόν, ο Χωσέ Μανουέλ Μαργκάγιο πρώτα έχει το λόγο γιατί ξέρω ότι θέλει να θέσει ένα ερώτημα και μόλις του απαντηθεί να μας πει τι γίνεται και με τα θέματα της εποπτείας. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον Επίτροπο. Είσαστε ο πρώτος που αναλαμβάνει τόσο υψηλές ευθύνες εντός των θεσμικών οργάνων της Ένωσης και να έρχεται εδώ μπροστά μας να μιλήσει μετά από τα όσα έγιναν με την Ελλάδα. Δεν θα επικεντρωθώ πάλι στην Ελλάδα, απλώς η κατάσταση με την Ελλάδα δείχνει, όπως είπαν πολλοί, ότι αυτή είναι η πρώτη ημέρα της ζωής του ευρώ. Καταρχήν πρέπει να προχωρήσουμε μέσα σε μια καταιγίδα και να δούμε πώς θα καταλήξουμε σε ήρεμα νερά. Τα πράγματα όμως είναι πολύ διαφορετικά όταν προσπαθεί κανείς να πλοηγήσει το καράβι του μέσα σε μια καταγίδα. Τώρα, στο τομέα της περιπτωσιολογίας είδαμε ότι υπάρχουν κάποια, α, κάποια αντιφατικά κάποιες αντιφατικές δηλώσεις από τον πρόεδρο του, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας που είπε ότι δεν θέλει να εμπλακεί το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο γιατί αυτό θα σήμαινε ότι εκχωρούνται εξουσίες προς το Ταμείο και υπήρξε μια απόρρεψη της γενικής ιδέας ε, των κοινών, ε, έκδοσης κοινών ομολόγων ε, των χωρών της ζώνης του ευρώ για την χρηματοδότηση της, οικονομίας με πιο, της ελληνικής οικονομίας με πιο χαμηλά επιτόκια έτσι ώστε να μπορέσει να ενισχυθεί και η ανάπτυξη και η ανάταση της ελληνικής οικονομίας. από πλευρά προπολογισμού. Τώρα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα λέει ότι η έκδοση των ομολόγων θα πρέπει να απορριφθεί ω ιδέα γιατί θα πρέπει να ακολουθήσουμε το δόγμα ο πληρώνει. Ε, εντάξει, εγώ συμφωνώ μαζί σας ότι πρέπει όντω να δημιουργηθεί ένα ταμείο έτσι ώστε να μπορεί κανείς να συμβάλλει στην δική του σωτηρία από μόνο του. Τώρα, η ελληνική περίπτωση δείχνει ότι οι στατιστικές έχουν αποτύχει απόλυτα. Υπήρξαν κονδύλια και πιστώσεις που επιτρέψανε να καλοπιστούν τα δημοσιοοικονομικά της, Ευρω... της ελληνικής δημοκρατίας. Μήπως θα μπορέσουμε με το πακέτο αυτό που προτείνεται να υπάρξει κάποια βοήθεια ώστε να μην μπορεί να υπάρξει αυτή η διαδικασία και η δυνατότητα καμουφλαρίσματος των ελλημάτων. Όλα αυτά επίσης έγιναν και με μια συνεργασία απαραίτητη συνέργεια, όπως λέγεται στο δίκαιο, της ελληνικής κυβέρνησης με ορισμένε τράπεζες οι οποίες διευκόλυναν αυτές τις ενέργειες. Μήπως μια σωστή ευρωπαϊκή εποπτεία δεν επέτρεπε να γίνουν τέτοιου είδους ε, συνεργασίες και συνωμοσίες και θα ήταν χρήσιμο να έχουμε ενώπιόν μας τους Έλληνες ρυθμιστές να μας πει τι κάνανε όταν γινόντουσαν αυτές οι ενέργειες. Τρίτον, σε ό,τι αφορά τις χρηματοοικονομικές αγορές, είναι σαφές ότι η διάσωση δεν αφορά μονάχα την αγάπη μας για την Ελλάδα αλλά και την ανάγκη να διασωθούν ορισμένες τράπεζες στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι οποίες κατέχουν ελληνικά ομόλογα. Και το ερώτημά μου είναι, θεωρεί ο κύριος Επίτροπος απαραίτητο να απαγορεύσει ορισμένα προϊόντα τα οποία έχουν συμβάλει τα μάλα στην ε, κερδοσκοπία κατά της Ελλάδος, τα CDS παραγματικά τα... οι συμφωνίες ανταλλαγής κίνδυνου αθέτησης το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξάλλου προσπαθεί να προωθήσει στο βαθμό του δυνατού τα θέματα εποπτείας. Είναι το Συμβούλιο το οποίο έχει την πρώτη ευθύνη να προσπαθήσει να πλησιάσει στις θέσεις μας και ζητώ συγγνώμη γιατί πρέπει να αποχωρήσω, αλλά είμαι σίγουρος ότι θα καταγράψει ο συνεργάτης μου τα, τις απαντήσεις σας στα ερωτήματά μου. Um, Πρόεδρος, ευχαριστούμε πολύ. Είχαμε σύντομη εισαγωγή λοιπόν εκ μέρου του Αντιπροέδρου. Σα υπενθυμίζω, αν ο καθένα μιλήσει 3,5 λεπτά δεν θα έχουμε απαντήσει. Σα παρακαλώ λοιπόν συνάδελφοι, κρατηθείτε μέσα στο ένα λεπτό. Ζαν Πολ Να σα διαβάσω τα ονόματα. I've Gauzes, Vertman-Kool, Beres, Jury, Lamberts, Clint, Swinburne, McCarthy, Podimarty, Oconee, Hockmark, Ford, Dominici, Clute, Bullman, and I'm sure there's somebody I've missed. Σίγουρα κάποιον θα ξέχασα. Κάμφεν. Άλλος. Κλείνει ο κατάλογος αυτή τη στιγμή. Ζαν Πολ Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επιτροπέ. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που είστε εδώ μαζί μας και σημειώνουμε την αποφασιστικότητά σας, τη σαφήνεια του προγράμματός σας και την πραγματική βούληση να βελτιωθεί η λειτουργία όλων όσων έχουν σχέση με τα χρηματοπιστωτικά. Μας το είπατε, έχετε αρχίσει να το κάνετε. Οι υπηρεσίε σας δουλεύουν πολύ συντονισμένα για το πρόγραμμα αυτό. Δύο παρατηρήσει τώρα. Καταρχήν το IFM που δεν αφορά που αφορά Γενικότερα όλα τα ταμεία που δίνουν είναι στο ΠΣΕΒΕΜ. Το Κοινοβούλιο έχει προσφέρει μεγάλο έργο στην κατεύθυνση αυτή και οι συζητήσεις με τους κοιόδες με των άλλων ομάδων πήγανε πάρα πολύ καλά. Βέβαια δεν πρέπει να βιαζόμαστε και να προδικάζουμε καταστάσεις. Ελπίζω όμως ότι μεγάλη πλειοψηφία θα υποστηρίξει αυτό το πρόγραμμα που είναι αναγκαίο και η συζήτηση με το Συμβούλιο θα είναι σίγουρα δύσκολη. Θα επανέλθω σε αυτό που είπατε για τις ε, οργανισμούς αξιολόγησης. Υπήρξε εισηγητή στην προηγούμενη πενταετία του κανονισμού για τα, τους οργανισμούς αυτούς και σας ερωτώ, πείτε μας, πότε θα δημοσιεύσετε, θα κυκλοφορήσετε το κείμενο εφαρμογής, γιατί χρειάζονται δύο κείμενα. Ένα κείμενο για τη μεταβατική περίοδο, για την καταγραφή σε μητρό εποπτεία κλπ. Και ένα δεύτερο κείμενο που έχει σχέση με την χρηματοπιστωτική εποπτεία, το σχετικό με τις εξουσίες ελέγχου της Ευρωπαϊκής Αρχής. Διότι ήμασταν πρώτοι που πετύχαμε ότι η εποπτεία αυτών των οργανισμών αξιολόγησης να γίνεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και επιτρέψτε μου να σας δώσω και μια συμβουλή γνώμη. Στη δουλειά αυτή που γίνεται, μελέτης κλπ. Αναφέρθηκε και το θέμα της αξιολόγησης κρατών. Απάντηση κατάλληλη ακόμα δεν πήραμε. Επίσης αναφέρθηκε η δυνατότητα να υπάρξει ένα ευρωπαϊκός οργανισμός αξιολόγησης. Ακαθόδες θέμα. Αξίζει να μελετηθεί. Δεν νομίζω ότι υπάρχει μία μόνο λύση. Η πραγματικότητα είναι η αλήθεια. Δηλαδή πρέπει οι χρηματοπιστωτικές αγορές να καταλάβουν ότι οι οργανισμοί αξιολόγησης δεν μπορεί να είναι ο μόνος δείκτης, ο μόνος γκουρού. Πρέπει να είναι ένα κριτήριο μεταξύ πολλών προκειμένου να αξιολογηθεί η οικονομική πολιτική του κάθε κράτους. Ευχαριστώ. Πρόεδρος. Άφησε το Ζανπόλ να ξεπεράσει το ένα λεπτό γιατί στην προηγούμενη συζήτηση δεν χρησιμοποιεί το χρόνο του. Η κυρία Βάλμαν Κόχ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τον κύριο Επίτροπο και να τον υποστηρίξω στην προσέγγιση του όταν μας είπε ότι θέλει ένα πολύ συγκεκριμένο πακέτο ευρωπαϊκό όπως επίσης και στην προσπάθειά του όπου οι G20 προσπαθούν να κάνουν κάτι το οποίο να ισχύσει και για την Ευρώπη. Μόνο έτσι θα έχουμε λύση της κρίσης. Έχω όμως να κάνω μια ερώτηση. Σωστά προτείνεται ένα πολύ συγκεκριμένο πακέτο και για τις τράπεζες και για τις ασφάλειες προκειμένου να εξασφαλιστεί η σταθερότητά τους. Όμως το πακέτο αυτό έχει επιμέρους στοιχεία ψηφίδες του παζλ αυτού. Η φερεγγιότητα, η αποκατάσταση της έφραυσης ε, της οικονομίας, αλλά γίνουν αυτά, όλα αυτά οι τράπεζες πρέπει να, είναι στο ύψος της πρώτης τους ευθύνης, δηλαδή αρμοδιότητες του που να δίνουν πιστώσεις στη βιομηχανία. Πρέπει να μπορούν οι τράπεζες να ασκούν πλήρως αυτή τη δραστηριότητα. Ερωτώ λοιπόν, στις προτάσεις σας θα κάνετε συνολική αξιολόγηση όλων αυτών των στοιχείων ψηφίδων του παζλ. Δεύτερο, μια δεύτερη ερώτηση για το ε, IFM και τις τρίτες χώρες. Σωστά αναφερθήκατε στη σημασία εφαρμογής στο πλαίσιο των G20. Έχω την αίσθηση ότι στο συμβασμό που προτείνεται και είχαμε πρόσθετες δηλώσεις του Υπουργού Σόιμπλε και της Υπουργού Λαγκάρντα Ποια είναι η γνώμη σας για τα συνταξιοδοτικά ταμεία, για το private equity και δεν θέλω να μιλήσω για τα hedge funds. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Επαναλαμβάνω, κρατηθείτε μέσα σε ένα λεπτό. Περβάως. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Πίτροπε για την εισαγωγή. Σας αναφερθήκατε σε εργασίες των G20. Βέβαια, δεν πρέπει να επικρίνουμε τους πάντες και τα πάντα, μόνο να αναγνωρίζετε όταν δείτε τα πορίσματα των G20, το πώς εφαρμόζονται εδώ ή εκεί. Καλύτερα θα ήταν να είχα μια διεθνή οργάνωση που να ετοιμάσει ένα κείμενο που να μην είναι καθαρά διακυβερνητικό, να υφίσταται πίεση από επιμέρους κράτη-μέλη και η Ένωση δεν θα πρέπει να εγκαταλείψει ένα τέτοιο όραμα αμοιβαιότητας. Τώρα, για, την, για το ελληνικό ζήτημα είπατε ότι η Ένωση προσπαθεί να βρει μέσω αλληλεγγύης και καιρό ήταν να γίνει αυτό. Δεν ξέρω αν είστε ικανοποιημένοι με αυτό που έγινε το Σαββατοκύριακο, το πώς διαχειρίστηκε η Ένωση την κρίση αυτή. Εγώ προσωπικά δεν ε, είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένη και καλό θα είναι να τα λέμε αυτά. Ε, θα ήθελα να κάνω ένα διάλογο με τον Σάφο Γκοζές μπροστά σα για του οργανισμού αξιολόγηση. Ήταν όντω εισηγητή. Πιστεύω ότι το θέμα αυτό πρέπει να συνεχίσουμε να το μελετάμε. Τέθη το θεωρητικό ερώτημα. Όλα τα προϊόντα που βαθμολογούν η και αυτοί είναι στο ίδιο επίπεδο. Το κρατικό χρέο είναι διαφορετικό. Έπειτα η ευθύνη, η στανταρ μου της είναι υπόλογο σε ποιον για τη βαθμολόγηση που δίνει. Σε ποιον είναι υπόλογος. Το θέμα λοιπόν της ευθύνη και τις υπολογίες αυτή ακόμα δεν έχει μελετηθεί σε βάθος. Και ένα τελευταίο το πιο σημαντικό θέμα, κύριε Επίτροπε. Αν δούμε τις αιτίες αυτής της κρίσης, έχουν σχέση με συμφέροντα, με υπερβολικές ωρέξεις, αλλά και με θέματα κανονισμού. Δηλαδή οι κατασκευαστές των προϊόντων, τραπεζικών προϊόντων και οι επόπτες από τη μεριά τους απείλησαν ότι θα εγκαταλείψουν μια χώρα αν ασκηθεί μια ρύθμιση και τελικά η ρύθμιση από ορισμένου μεγάλους φορείς και δεν θέλω να αναφέρω ονόματα πρώτες και καλύτερες οι μεγάλες τράπεζες επενδύσεων και ρωτώ τι άλλαξε σήμερα και συνεχίζεται αυτό επιτρέψτε μου κύριε Πρόεδρε στην Επιτροπή της Βασιλείας γιατί ακούμε άλλες φορές εκεί πέραν από αυτούς που ρυθμίζουν τις τράπεζες. Δηλαδή τι θέλω να πω. Γιατί δεν βάζετε παράγγελα και τις προτάσεις του Ευρωκοινοβουλίου να υπάρξει μια γραμμή στον προπολογισμό ειδικά για την εμπειρογνωμοσύνη. Πέραν αυτών των μεγάλων λόμπι των τραπεζών και των υποπτικών οργάνων, στο προηγούμενο ε, Κοινοβούλιο ψηφίσαμε ένα κείμενο. Γιατί δεν είναι μόνο η, θέμα, η σταθερότητα της τράπεζας, είναι και η χρησιμότητα της τράπεζας για το όλο σύστημα. Πρόεδρος, αγαπητοί συνάδελφοι, κοιτάξτε. Όλοι οι συνάδελφοι, από ό,τι φαίνεται, θέλουν να κάνουν σχόλια και όχι να ακούσουν απαντήσεις. Αν στο τέλος δεν υπάρχει χρόνος για απαντήσεις, θα ζητήσουμε από τον Επίτροπο να μας απαντήσει γραπτά. Άλλη λύση δεν υπάρχει αν ο καθένας μιλάει δύο και τρία λεπτά. Η κυρία Τζούρι. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ κατάγομαι από μια χώρα που θα αναλάβει την Προεδρία του Συμβουλίου, από την Ουγγαρία, και θα ήθελα να μάθω ποια ακριβώς θα είναι τα καθήκοντα κυρίως για το θέμα 3 και, για το τρίτο και τέταρτο θέμα που αναφέρατε για τις οδηγίες ε, για τα equities. Υπάρχει και ένα ε, χρονοδιάγραμμα G20 και ε, υπάρχει το CRD 3 και 4. Υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα της G20 και υπάρχει και ένα ευρωπαϊκό χρονοδιάγραμμα. Η Κομισιόν ποιο ακριβώς χρονοδιάγραμμα έχει. Πώς θα τα συνδυάσετε τα δύο χρονοδιαγράμματα γιατί αλλιώ θα υπάρξει πρόβλημα και για τις τράπεζες και για τις επιχειρήσεις και για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις κυρίως που δεν θα μπορούν να δανειστούν. Οι ΙΠΑ ακόμη δεν έχουν πληρώσει τα της Βασιλείας 2, οπότε πώς θα αποφύγουμε τον, την οποιαδήποτε στρέβλωση του ανταγωνισμού. Ξέρω ότι γίνονται κάποιες αξιολογήσεις επιπτώσεων τώρα αλλά θα πρέπει να υπάρξει μια διαφοροποίηση. Γι' αυτό ρωτώ. Οι ε, μελέτες επιπτώσεων πόσο έχουν προχωρήσει. Ευχαριστώ. Ο Φιλίπ. Yes, Actually, I'm a bit... Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ήθελα να ακούσω απαντήσεις από τον Επίτροπο όμως. Για την περίπτωση της Ελλάδος, λοιπόν, νομίζω ότι έδειξαν οι ηγέτες της Ευρώπης στα, τους τελευταίους πέντε μήνες μια έλλειψη πνεύματος ευθύνης και έλλειψη αλληλεγγύης αν έχει οξυνθεί η κρίση είναι ακριβώς λόγω της απραξίας της Ευρώπης. Το ερώτημά μου δεν έχει να κάνει με την Ελλάδα, το θέμα έχει να κάνει με τα επιτρεπόμενα εργαλεία και πρακτικές. Είναι κάτι που συζητήσαμε χθε σε σχέση με την οδηγία κεφαλογικής Επαρκίας 4, σε 4. Ποια είναι η αποψή σας προσωπικά σε σχέση με το να χωριστούν οι τραπεζικές δραστηριότητες, που είναι μια λύση για αυτό το πρόβλημα, να ξαναδιαχωριστούν οι τράπεζες νομικά, να υπάρχουν είτε να διαλυθούν οι τράπεζες οι οποίες κάνουν και τα δύο αυτά, είτε να υπάρξουν κάποια α, φράγματα μεταξύ των κεφαλαίων των τραπεζών που είναι επενδυτικές τράπεζες και των τραπεζών που λειτουργούν με καταθέτες και δάνεια. Αυτά, σε ένα λεπτό μονάχα. Right, the commissioner wants to try and come... Η Κομισιόν θα προσπαθήσει να επανέλθει σε μερικά από τα θέματα αυτά. Θα προσπαθήσω. Σας ζητώ συγγνώμη γιατί μερικές φορές είμαι κάπως ε, τηλεγραφικού χαρακτήρα. Προσπαθώ να απαντήσω λοιπόν στα πρώτα ερωτήματα που μου ετέθηκαν και σας ευχαριστώ για τις παρεμβάσεις. Σφαίρα εφαρμογής καταρχήν αχανής. Σε ό,τι αφορά για την οδηγία EFM, ο στόχος της και η σημασία της είναι να καλύψει με ένα αποτελεσματικό και ισορροπημένο τρόπο, γιατί αφορά πολλούς φορείς, πολλού, πολλά ευρήματα, διαφορετικά είδη κεφαλαίων. Διευκρινίζοντας και διαφοροποιώντας, και αυτό είναι το αντικείμενο ενδελεχούς προσπάθειας της Κομισιόν, να γίνει αυτή η διαφοροποίηση με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Αυτό σας είπα εξάλλου Γι' αυτό το θεμελιώδες θέμα για το οποίο εγώ θέλω να φέρω διαφορετικέ προτάσεις τον Ιούνιο ή τον Ιούλιο για τα παράγωγα. Είπαμε ότι θα διαφοροποιήσουμε στην αντιμετώπιση μας μεταξύ των χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων και των επιχειρήσεων που είναι βιομηχανικού χαρακτήρα, οι οποίες χρησιμοποιούν κάποια από αυτά τα προϊόντα για αντιστάθμιση κινδύνου. Ξέρω λοιπόν κυρία Πρόεδρε ότι πρέπει να δούμε όλα αυτά τα πράγματα προσεκτικά επί τη βάση της φύσης της δραστηριότητας κάθε παίκτη στις αγορές. Κύριε Γκασία Μαργκάγιο, ο οποίος μου εξήγησε ότι έπρεπε να φύγει, αναφέρθηκε στην ελληνική κρίση. Κύριε Λαμπέρ, δεν ήμουν αισιόδοξο. Και όταν μιλάμε για την αισιοδοξία θυμάμαι το Ζαν Μονέ που λέει δεν είμαι ούτε αισιόδοξο ούτε απεσιόδοξο, είμαι αποφασισμένος. Δεν είμαι λοιπόν αισιόδοξο ούτε νιώθω εφορία σε σχέση με τον τρόπο που διαχειριστήκαμε στην πράξη την ελληνική κρίση. Δεν θα επανέλθω σε αυτά τα οποία έγιναν από τον συναδελφό μου τον κύριο Όλη Ρέν, ο οποίος θα σας εξηγήσει ο ίδιος το ρόλο που διαδραμάτισε η Κομισιόν. Αλλά υπάρχουν δύο θέματα για τα οποία ως υπεύθυνο επίτροπος για την εσωτερική αγορά και τις υπηρεσίες ενεκλήθην και θα πρέπει να παρέμβω αφορά καταρχήν το ένα θέμα τις κινήσεις στην αγορά ορισμένων ειδών προϊόντων, ιδίως των ε, σέδες των συμβολέων ανταλλαγής αθέτησης για το δημόσιο χρέος και επίσης υπάρχει το πρόβλημα των αρμοδιοτήτων και της κατανομής των κατοικών. Ποιος κάνει τι. Όλα αυτά τα οποία έχουν γίνει με κάνουν να πιστεύω ότι απαιτείται μια πλήρης ρύθμιση όλων των παραγόγων προϊόντων με την υποχρέωση συμψηφισμού και εγγραφής σε trade repositories, σε μητρώα συναλλαγών. Αυτό λοιπόν θα αποτελέσει αντικείμενο προτάσεων που θα διατυπωθούν ήδη το καλοκαίρι. Και οι Αμερικανοί νομίζω, θα δω και την επόμενη εβδομάδα, αλλά νομίζω ότι έχουν ήδη κάποια προπορία απέναντί μας για τα θέματα αυτά ρύθμισης. Αυτό είναι ο πρώτο τομέα, το πώ θα χρησιμοποιήσουμε τα διδάγματα τη κρίση. Το δεύτερο αφορά του φορεί πιστοποιητική αξιολόγηση που αναφέρθηκαν από εσά, που έχουν μια μεγάλη εξουσία αυτή η φορείς. Και για τις επιχειρήσεις, για τα προϊόντα τα χρηματοπιστωτικά, αλλά και έναντι των κρατών. Γι' αυτό εγώ ζήτησα να υπάρχει μεγαλύτερη ευθύνη από τους φορείς αυτούς και υπενθύμησα στον κύριο Κοζές το χρονοδιάγραμμα ότι θα πρέπει από τις 7 Ιουνίου να υποβάλλονται αιτήσει καταγραφής αυτών των φορέων εγώ θα κοιτάξω τα κείμενα αυτά για να δούμε αν είναι επαρκή προδιαγραφέ ή όχι και η πρόθεσή μα είναι να είναι το νομοθέτημα αυτό λειτουργικό ήδη από το Δεκέμβριο. Επέκεινα όμω πρέπει να πάμε μακρύτερα να δούμε ποιο είναι ο αντίκτυπο αυτή τη αξιολόγηση στο σύνολο του χρηματοπιστωτικού συστήματο, ακόμα και του οικονομικού συστήματο. Γι' αυτό θα πρέπει να σκεφτώ. Χωρί όμω να αυτοσχεδιάσω, για να αντιμετωπίσουμε και την απαραίτητη πολυμορφία και τον ανταγωνισμό σε αυτόν τον τομέα που αυτή τη στιγμή έχει ε, ουσιαστικά δεσπόζεται από τρεις μεγάλες εταιρείες. Ένα άλλο στοιχείο είναι η σύγκρουση συμφερόντων. Το κείμενο το οποίο θα σας ε, υποβληθεί το Δεκέμβριο αντιμετωπίζει το θέμα αυτό. Θέλουμε να δούμε αν θα είναι αποτελεσματικό ή επαρκές. Θα το επεξεργαστούμε και τις επόμενες ημέρες για τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού φορέα δεν μπορώ να σας πω αν θα είναι δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου, αν θα είναι ανάμεικτου δικαίου ή ιδιωτικού δημοσίου. Δεν μπορώ να σας πω ότι θα είναι ένας φορέας ειδικό για το έργο αυτό, την ανάλυση των κινδύνων που έχουν να κάνουν με το κρατικό χρέος, ή γενικότερος φορέας, αλλά σίγουρα χρειάζεται να υπάρχει και ένας ιδιαίτερος φορέας για να εξασφαλίσει μια μεγαλύτερη αντικειμενικότητα στον τομέα αυτό. Αυτά είναι τα δύο διδάγματα τα οποία μπορούμε να λύσουμε. Αν μου επιτρέπετε, κυρία Πρόεδρε, υπάρχουν και άλλα γενικότερα συμπεράσματα από την κρίση ό,τι αφορά την ευκυβερνησία της ευρωπαϊκής οικονομίας και είμαστε μακρά ακόμα από το να επιτύχουμε τους στόχους μας σε ό,τι αφορά την απαραίτητη μορφή συντονισμού των οικονομικών και δημοσιονομικών πολιτικών σε ευρωπαϊκή, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στη ζώνη του ευρώ. Θα πρέπει λοιπόν να εξασφαλίσουμε και την αξιοπιστία των στατιστικών στοιχείων, γιατί εκεί φάνηκε ότι πραγματικά είχαμε μεγάλες ελλείψεις. Ίσως. Ίσως. Μπορώ να απαντήσω και πάλι πιο τηλεγραφικά. Στην κυρία Βότμα Κολ, αναφερθήκατε στην ανάγκη μιας συνολικής προσέγγισης Γι' αυτό πάω στι ΗΠΑ. Το ίδιο θα κάνω και στην Κίνα και σε άλλε περιοχέ του κόσμου. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτό που είπα, η τριπλή, ε, τριπλή προσαρμογή. Ξέρουμε ότι τα δύο τρίτα των επιχειρήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση χρηματοδοτούνται από τις τράπεζες. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και λέω ναι στο θέμα της αξιολόγησης που εμείς θα εξετάσουμε πάρα πολύ προσεκτικά για τα συνολικά, τα μελλοντικά μέτρα ρύθμιση στον τομέα των τραπεζικών σε ό,τι αφορά την δάνειο λυπτική ικανότητα. Η κυρία Μπερέσα αναφέρθηκε στους G20, καλύτερα 20 παρά 7 ή 8 και εκεί θα πρέπει να βελτιώσουμε την παγκόσμια ευκυβερνησία στον χρηματοοικονομικό τομέα. Είναι ένα θέμα το οποίο με ενδιαφέρει πάρα πολύ, το θέμα της τροφιμικής ασφάλειας. Επίσης και εκεί θα πρέπει να έχουμε καλύτερη διακυβέρνηση. Χρειαζόμαστε, αυτό φαίνεται από την κρίση, να έχουμε εργαλεία οικονομικά, νομισματικά και χρηματοοικονομικά. Αυτό επομένως θα με οδηγήσει μέχρι την επόμενη άνοιξη να προσπαθήσω να συμπληρώσω αυτή την εργαλειοθήκη εργαλείων για την, το χρηματοοικονομικό στίβο, για τους φορείς πιστοληπτικής αξιολόγησης θα πρέπει να έχουν μια ευθύνη όταν κάνουν οικονομικές αναλύσεις, να βασίζονται μεν στα στοιχεία τα οποία παρουσιάζει μια χώρα σε επίπεδο προπολογισμού και οικονομία, αλλά να ξέρουν και ποιε είναι οι αιτίε όλων αυτών, να δουν ποια είναι τα, οι πηγές αυτών των προβλημάτων. Στην Ελλάδα υπήρξε μια απότομη επιδείνωση, αλλά θα πρέπει οι φορεί να βλέπουν τη χώρα αυτή στο πλαίσιο το πλήρε τη, να τη βλέπουν σε βάθο χρόνου, όχι απλώ να την αξιολογούν επειδή είναι μέλος της ζώνης του, του ευρώ, αλλά να τη βλέπουν σαν συνολικό οικονομικό γίγνεσθε. Και εγώ εμποδίζομαι να απαντήσω σε όλα αυτά, αλλά θα επανέλθω σε αυτά τα θέματα. Λοιπόν, κοιτάξτε. Το ρολόι αυτό βράδυ βραδιπορεί. Έχουμε μισή ώρα και μέσα στη μισή αυτή ώρα έχουμε δέκα και περαιτέρω ομιλητές. Όλοι θα μιλήσετε. Αλλά στο ένα λεπτό θα σας αποκόψω το λόγο ως άλλη προκρούστρια. Και πραγματικά δεν θέλω να σας περιορίσω ούτε εσένα, Βολφ, που είσαι ο επόμενος. Ευχαριστώ. Κύριε Επίτροπε, μιλήσατε για ένα ταμείο για να μπορούμε να αποκαταστήσουμε κάποιους ε, δομέ, κάποιες τέτοιες ζημιές στο μέλλον. Δεν είναι απόλυτα σαφές. Πώς ακριβώς θα βοηθήσει αυτό το ταμείο και μας ε, είπατε ότι θα επιβαρυνθούν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που μέχρι, μέχρι τώρα δεν είχαν σχέση με την ε, κρίση. Τι ακριβώς εννοείται. Τώρα, δεν θα έπρεπε να υπάρξουν ε, στρεβλώσεις στον ε, ανταγωνισμό και επίσης οι εταιρείε private equity νομίζω είναι επιπισμένες και αποτελούν ένα κομμάτι της χρηματοδότησης όλων αυτών των ταμείων. Ο Μάριο Μόντι επίσης υποβάλλει μια έκθεση για την εσωτερική αγορά και την ενίσχυσή τη. Τι ακριβώς περιμένετε εσεί από αυτή την έκθεση και θέλετε να προσθέσετε κάτι στην έκθεση αυτή. Ευχαριστώ. Ωραία. Ακολουθήστε το παράδειγμα όλοι του Βολφ. Ε, ευχαριστώ Πρόεδρε. Χαίρομαι που έχετε αφοσιωθεί τόσο πολύ στο έργο σας για την καλύτερη δικυβέρνηση και την αντιμετώπιση των προβλημάτων και για τις ε, χρηματοοικονομικές υπηρεσίες. Το θέμα όμως που θα έχετε να αντιμετωπίσετε με την μετάβαση για, το, ε, για την ε, διακυβέρνηση. Δεν πρέπει να έχουμε πιο συντονισμένο τρόπο για να δούμε όλες τις προτάσεις που υπάρχουν και τις επιπτώσεις που θα έχουν στην χρηματοδότηση της πραγματικής αγοράς. Υπάρχουν κάποιοι τομείς που θα ήθελα να τους τονίσω. Ας πούμε, για τα παράγωγα. Αν θέλουμε να δούμε εξαιρέσεις, ε, τότε θα πρέπει σίγουρα να δούμε και κάποια είδη εξαιρέσεων. Ας πούμε για την, ε, για τα, για την ε, νομοθεσία του CRD που θα πρέπει να αφορά τις, τη χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων. Ε, θα μου πείτε ποιες είναι οι απόψεις γι' αυτό. Ευχαριστώ. Κάποιος μου κλέβει τον κατάλογο. Δύο σχόλια. Επικεντρωνόμαστε στη διαφάνεια, Επίτροπε. Μήπως πρόκειται να υποβάλλετε οποιαδήποτε α, πρόταση για τις σκοτεινές δεξαμενές και πώς πρόκειται να ρυθμίσετε τις τράπεζες οι οποίες κρύβουν τα δημόσια χρέη και επίσης όταν θα μιλήσετε στις ΕΠΑ μπορείτε να πείσετε τη είπα, να ε, επιταχύνουν το, τις δραστηριότητες τους για το CRD3 και να μην έχουμε καθυστερήσεις και να έχουμε έγκαιρο χρονοδιάγραμμα, έγκαιρη εφαρμογή έτσι ώστε να μπορέσουν να υπάρξουν τα αποθυματικά των τραπεζών. Ευχαριστώ. Ε, Η Άννη Ποδήματα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Τηλεγραφικά, ε, κύριε Επίτροπε, ευχαριστώ πολύ καταρχήν για την ε, εισαγωγική σας παρέμβαση και για τις εξαιρετικές απαντήσεις σας. Σε σχέση με τα ε, ασφάλιστρα κινδύνου επικρατικών ομολόγων, ένα ερώτημα. Είναι προφανές ότι σε ό,τι αφορά την ελληνική περίπτωση τα CDS, τα ασφάλιστρα κινδύνου των ελληνικών κρατικών ομολόγων δεν ευθύνονται για τη δημιουργία του προβλήματος, αλλά είναι επίσης προφανές ότι έχουν παίξει σημαντικό ρόλο στην επιδείνωση της κατάστασης της ελληνικής οικονομίας, στην επιβάρυνση του ελληνικού δημόσιου χρέους και τη διεύνηση του δημοσιονομικού ελλείμματος. Επειδή σε συνέχεια της ε, επιστολής των τεσσάρων πριν από μερικές εβδομάδες αναλάβατε να διεξάγετε μία έρευνα για το ρόλο των CDS στην αγορά κρατικών ομολόγων. Ήθελα να σας ρωτήσω, σεβόμενοι ότι δεν μπορείτε να μας δώσετε λεπτομέρειες, ποια είναι τα βασικά συμπεράσματα στα οποία έχετε οδηγηθεί μέχρι σήμερα σε ό,τι αφορά τον ρόλο των, των CDS στην επιδείνωση της ελληνικής κρίσης και το δεύτερο σε ό,τι αφορά τους διεθνούς οίκους πιστοληπτικής αξιολόγησης. Ε, συμφωνώ απολύτως με αυτό που είπατε κύριε Επίτροπε, ότι θα είναι μια λύση να δημιουργηθεί ένας ευρωπαϊκός οίκος αξιολόγησης, καθότι δεν είναι ζήτημα απλώς μεγαλύτερης διαφάνειας, θεωρώ ότι είναι ζήτημα δημοκρατίας και εθνικής κυριαρχίας και θέλω να σας ρωτήσω πώς αυτή την πτυχή σκοπεύετε να την αντιμετωπίσετε. Thank you. Um, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, καλημέρα σας. Αγαπητοί συνάδελφοι, όπως και εσείς και εγώ θεωρώ ότι θα πρέπει να έχουμε μεγαλύτερη σταθερότητα του τραπεζικού συστήματος, να αποφύγουμε την επιστροφή υπερβολικών κινδύνων με συγκεκριμένα εργαλεία διαχείρισης και ελέγχου. Και σχετικά με αυτό κύριε Επίτροπε, θα ήθελα να σας ρωτήσω για τα τοξικά στοιχεία ενεργητικού που ήταν στην αρχή της ως αιτία αυτή της κρίσης που μετά έγινε οικονομική και χρηματοπιστωτική. Αυτά τα τοξικά προϊόντα, ζητείτε να απαλλαγούν οι τράπεζε από τα, από τα τοξικά αυτά προϊόντα. Πώς θα γίνει αυτό, υπάρχει έλεγχος, τι γίνεται με αυτά. Δεύτερο, για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που εξακολουθούν να έχουν μεγάλες δυσκολίες για πρόσβαση σε δάνεια και πιστώσεις, ενώ οι τράπεζες εξακολουθούν να κερδοφορούν. Γιατί η Γαλλία τουλάχιστον Σήμερα 11 δις κέρδη έχουν οι τράπεζες. Δεν υπάρχει τρόπος να βελτιωθεί η πρόσβαση σε πιστώσεις των μικρομεσαίων μεσαίων επιχειρήσεων με δικές σας ενέργειες. Πρόεδρος. Κούνα. Ευχαριστώ. Για τις επενδύσεις που χρειαζόμαστε στην Ευρώπη θα δίσταζα να πω ότι ο χρηματοπιστωτικός τομέας ρηπαίνει και θα δίσταζα για την κρίση να πω ότι γενικά οι τράπεζες έχουν μειωμένα η ελληπή κεφάλαια. Διάβασα στο Financial Times σήμερα ότι ο πρόεδρος της Επιτροπής της Βασιλείας Νοτβαλίνκ δήλωσε ότι η επίπτωση των νέων απαιτήσεων και όρων μπορεί να σημαίνει μείωση οικονομικής ανάπτυξης κατά 1%. Ένας άλλος σχολιαστής είπε ίσως είναι παραπάνω από 1%. Όποιο και να είναι το νούμερο, είναι σωστό το ότι το αποτέλεσμα θα είναι λίγο παραπάνω στην Ευρώπη για διάφορους λόγους. Κύριε Πίτροπε, λοιπόν, διερωτώ με πώς θα πρέπει να κινηθούμε για να έχουμε μια αξιολόγηση για τους νέους κανόνες για το τραπεζικό σύστημα, πώς αυτό θα επηρεάσει τη σταθερότητα όλης της οικονομίας μας. Ευχαριστώ. Η δική. Η ερώτηση μου αναφέρεται στο τι θα κάνετε για τις συγκεκριμένες αιτίες αυτής της κρίσης, δηλαδή τοξικά, το, τοξικές τιτλοϊοποίησεις, επειδή οι τράπεζες έχουν μειωμένα κεφάλαια, γι' αυτό οι τράπεζες πρέπει να τις υποστηρίξουν. Και δεν το είδα αυτό ψηλά στις προτεραιότητες. Η 3 θα εισάγει νέους κανόνες κεφαλαίων. Για τις δραστηριότητες για τη Βασιλεία χθε ακούσαμε ότι από τις αρχές του χρόνου κάτι γίνεται. Μερικές, μερικοί όμως έχουν κάνει τροπολογίες με καθυστέρηση που θα φτάσει ενδεχομένω το 2013-2014. Ξέρω ότι χρειαζόμαστε μελέτη αξιολόγηση και επιπτώσεων και για όλο τον κόσμο. Δεν συμφωνείτε όμω, κύριε Πίτροπο, ότι είναι τελείω απαράδεκτο να περιμένουμε 5 και 6 χρόνια μετά το Lehman Brothers για να εφαρμοστούν κανόνε για τα συγκεκριμένα αυτά προϊόντα τα οποία δημιούργησαν την κρίση. Ο κύριο Ντομινίτσι. Καλημέρα κύριε Επίτροπε. Σας εύχομαι καλή δουλειά. Μας αναφέρετε ένα κείμενο για τα παράγωγα. Και σας ερωτώ, το κείμενο αυτό θα έχει ένα συγκεκριμένο κεφάλαιο για τα credit default shops, για τις ιδέες και πιο συγκεκριμένα σχέση μεταξύ αυτών των προϊόντων και του κρατικού χρέους. Και αν ναι, θα προτείνετε απαγόρευση αυτών των CDS γυμνών, δηλαδή αυτά που δεν αναφέρονται άμεσα στο συγκεκριμένο χρέος με το οποίο υποτίθεται είναι συνδεδεμένα, προσφέρουν δηλαδή την ασφάλεια. Ο Γιούργεν Κλούτ. Ευχαριστώ πολύ. Και η δική μου πολιτική ομάδα θέλει να σας ευχαριστήσει για το έργο σας. Έχω κάτι να πω όμως για του φορεί πιστοληπτική αξιολόγηση. Έχουμε αναφερθεί στην περίπτωση της Ελλάδος, αλλά και η Πορτογαλία και η Ισπανία έχουν να αντιμετωπίσουν ένα αμφιλεγόμενο ρόλο των πιστοληπτικών φορέων αξιολόγηση. Πραγματικά, είναι αυτή η δυνατότητα, είναι δυνατόν να αντιμετωπίζουμε τα κράτη σαν ένα απλώ επιχειρήσει. Ένα κράτο για μένα δεν είναι κάτι το οποίο μπορούμε να το συγκρίνουμε με μια επιχείρηση προσδιάση. Έχει άλλου ρόλου, έχει άλλη λειτουργία και γι' αυτό το ερώτημά μου είναι κάτι το οποίο έχει νόημα να υπάρχουν ε, πιστοληπτικέ αξιολογήσει των κρατών μελών και των κρατικών ομολόγων. Ευχαριστώ, ο Ούντο. Κύριε Επίτροπε. κάθε επιτυχία στο έργο σας και σας ευχαριστώ για την αποφασιστική σας προσέγγιση. Έχω να θέσω δύο ερώτηματα. Ο κ. Ντομινίτσι έχει αναφερθεί ήδη στα CDS. Κανείς δεν έχει καταφέρει να μας εξηγήσει γιατί χρειάζεται η δυνατότητα αγοράς συμβολέων ανταλλαγής ε, συμβολέων αθέτησης για κρατικά ομόλογα όταν δεν τα κατέχει ο ίδιος αυτά τα ομόλογα. Εδώ πρέπει να υπάρξει κάποια δράση των αρχών της Ευρώπης για να αντιμετωπιστεί αυτό το ερώτημα. Δεύτερο σημείο, χθε είχαμε μια ενδιαφέρουσα ε, ακρόαση σε σχέση με την ε, Οδηγία Κεφαλογικής Επάρκειας 4, την έκθεση του κ. Ότμαρ Κάρας, και φάνηκε ότι οι κανόνες όπως προβλέπονται στη Βασιλεία 3 δεν είναι προσαρμοσμένε στις ανάγκε των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Και υπάρχουν μεγάλα προβλήματα, θα υπάρξουν μεγάλα προβλήματα για τι εταιρείε για τις τράπεζες οι οποίε παρέχουν δανειοδότηση στις μικρομεσαίες επιχειρήσει. Θα υποστηρίξει εδώ η Κομισιόν και το Κοινοβούλιο για να μπορέσουμε να φτάσουμε σε νέε συμφωνίε οι οποίε θα υποστηρίξουν καλύτερα την οικονομία από ό,τι μέχρι τώρα. Και νομίζουμε ότι όλα αυτά τα οποία έχουν αποφασιστεί μέχρι τώρα δεν είναι επαρκή προ την κατεύθυνση αυτή. Ο Πασκάλ Καντέν. Κύριε Μπαρνία, καλημέρα σα, Σε λίγε μέρε θα πάτε στι ΗΠΑ και προφανώ θα μιλήσετε για παράγωγα προϊόντα εκεί. Εγώ θα ήθελα να ξέρω τι θα πείτε στου ομολόγου σα, στου Αμερικανού. Ε, σε σχέση με την ανάγκη να υπάρχουν ε, κεντρικοί φορεί συμψηφισμού στην περιοχή του ευρώ σε σχέση με τη διαλειτουργικότητα των συμψηφιστικών φορέων. Κατά πόσο εσεί θα υποστηρίξετε λοιπόν αυτήν την ιδέα τη διαλειτουργικότητα και κατά πόσο θα είσαστε υπέρμαχος του οι φορείς αυτοί συμψηφισμού στη ζώνη του ευρώ να μπορούν να έχουν ε, εποπτεία, να, να, καλύπτουν μάλλον όλα τα προϊόντα, τα παράγωγα τα οποία διακινούνται στον στο, στη ζώνη του ευρώ. Ευχαριστώ πολύ λέει η Πρόεδρος. Υπήρξε κάποια επικάλυψη στα διάφορα ερωτήματα τα οποία τέθηκαν. Εγώ θα ήθελα απλώς να προσθέσω στο τέλος το ότι εσείς κύριε Επίτροπε στην εισαγωγή σας είπατε και αυτό αφορά πολλά θέματα εποπτείας είναι γεγονός ότι περιμένουν πολλοί αδειμόνως την απάντηση που θα δώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και υπάρχουν πολλές συζητήσεις για το ποιος βρίσκεται πίσω από την κρίση, αν ήταν απλώ η σύγκληση πολλών φαινομένων και η συμβολή πολλών. Ξέρουν πολλοί ότι οι τράπεζες έπαιξαν ένα προεξάρχοντα ρόλο στην κρίση αυτή, Επομένω, για να μπορέσουμε να δείξουμε ότι πράγματι πήραμε δράση για να ενισχύσουμε την ε, κεφαλουχική επάρκεια στις τράπεζες και ιδίω στον τομέα του χαρτοφυλακίου συναλλαγών των τραπεζών. Πιστεύω ότι η ρύθμιση του τραπεζικού τομέα πρέπει να είναι από τα πρώτα θέματα που θα αντιμετωπίσουμε. Συγγνώμη που είναι τόσα πολλά τα ερωτήματα που πρέπει να τα απαντήσετε όλα αυτά, αλλά έχετε όλο τον υπόλοιπο χρόνο. Θα χρησιμοποιήσω το χρόνο όσο μπορώ να απαντήσω στα ερωτήματα αυτά. Ε, έχουμε μια σημαντική ημερησία διάταξη το απόγευμα στο σώμα των επιτρόπων. Τρίτη, παρόλα αυτά, είναι έκτακτο αυτό. Θέλω να απαντήσω στην κυρία Τζουρί, η οποία αναφέρθηκε στα θέματα της αξιολόγησης και τα αποτελέσματα της οδηγίας για την κεφαλουχική επάρκεια. Εμείς προβλέπουμε μέχρι το τέλος του έτους, αρχές 2011, για την CRD4, την Οδηγία Κεφαλογικής Επάρκειας 4. την οδηγια κεφαλογικη επαρκεια 4 συνεχιζονται οι διαβουλεύσεις και εγώ είμαι πάρα πολύ προσεκτικός στο περιεχόμενο αυτών των διαβουλεύσεων. Δεν αυτοσχεδιάζουμε και δεν είναι μια τεχνητή διαβούλευση. Σήμερα το πρωί ξεκίνησα μια ε, δημόσια ακρόαση για τα θέματα ασφαλιστικών εταιριών και τόνισα το πνεύμα μέσα στο οποίο ξεκινάμε αυτήν την διαβούλευση για τη CRD4. Όπως είπατε κυρία Ντιούρι, η συζήτηση, ο διάλογο με τις ΗΠΑ είναι πάρα πολύ σημαντικό. πρέπει να είναι με, σε πνεύμα εμπιστοσύνη και χωρίς αφέλειε Από καμία από τι δύο πλευρές πρέπει το χρονοδιάγραμμα που αναφέρατε μεταξύ των ε, οδηγιών CRD και των αποφάσεων του G20 να τον το πιο συνεκτικό και να προσπαθήσουμε να εξασφαλίσουμε μια συνάφεια και μια συνεκτικότητα μεταξύ αυτού που κάνουν οι Αμερικανοί και αυτού που κάνουμε εμείς. Γι' αυτό εγώ θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η επίσκεψη στι Ηνωμένες όπως και στα άλλα μέρη του κόσμου γιατί ένα μεγάλο μέρος των αγορών είναι αμερικανικές και ευρωπαϊκές και δεν μπορούμε να τις παραγνωρίσουμε όπως δεν μπορούμε να παραγνωρίσουμε και τις ασιατικές αγορές εξάλλου. Κύριε Λάμπερτ, επανέρχομαι στο θέμα της, του διαχωρισμού των δραστηριοτήτων των τραπεζών. Κάτι μια ιδέα που ξεκινά από τις ΗΠΑ. Η ευρωπαϊκή τραπεζική δομή δεν είναι ίδια όπως η αμερικανική και η μορφή χρηματοδότηση οικονομίας μας δεν είναι ίδια στην Ευρώπη όπως στις ΗΠΑ. Η προσέγγιση της Κομισιόν δεν πηγαίνει προς την κατεύθυνση του διαχωρισμού των δραστηριοτήτων των τραπεζών, των τραπεζών, αλλά με δραστηριότητες μάλλον, αλλά στη συνολική εποπτεία των τραπεζών, ακόμα και αν έχουν διαφορετικές δραστηριότητες. Ο κ. Λαμπέρ έφυγε βέβαια, αλλά νομίζω ότι χρειάζεται μια διπλή εποπτεία. <clears throat> μια εσωτερική εποπτεία, που είναι θέμα διακυβέρνηση των επιχειρήσεων, στον πιστοτικό τομέα, και η κυρία Σουίμπον το έθεσε το θέμα αυτό, και από την άλλη πλευρά η εξωτερική εποπτεία από τις εθνικές ή ευρωπαϊκές αρχές. Χρειάζεται λοιπόν η διπλή εποπτεία για τον τραπεζικό τομέα και σας υπενθυμίζω ότι στην περίπτωση της Ευρώπης, ότι στις μισές από τις 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουμε σχεδόν τις μισές τράπεζες που ανήκουν σε εξωτερικούς φορείς, σε τράπεζες που είναι από το που η έδρα του είναι εκτό τη Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τουλάχιστον είναι εκτός της χώρας στην οποία βρίσκεται η τράπεζα και χρηματοδοτούν τα εκτό της ε, αγοράς αυτές οι τράπεζες. Λοιπόν, γι' αυτό χρειάζεται να υπάρχει διπλή εποπτεία. Ετέθηκε το θέμα της αγορας αυτες τι τράπεζε. λοιπον γι αυτο χρειαζεται να υπαρχει διπλη εποπτεια ετεθηκε το θεμα της εμπειρογνωμοσυνης για τα θέματα αυτά. Ε, αναφερθήκατε και σε μία γραμμή του προπολογισμού. Θέλω να σας υπενθυμίσω ότι η Κομισιόν δρά ως ανεξάρτητος εμπειρογνώμων. Και εγώ ορκίστηκα χθες ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, διότι είμαι υποχρεωμένος να το πράξω αυτό. Και το σύνολο των ε, ε, συνεργατών μου και αυτοί δρούν ως ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες. Και ήταν πάρα πολύ σημαντική αυτή η συζήτηση που έγινε και μας ε, είπαν ότι θα έπρεπε να δούμε αν χρειάζεται να υπάρχει μεγαλύτερη υποστήριξη του ESB σε ευρωπαϊκό επίπεδο. ώστε να βοηθήσει και τους χρήστες αυτών των ε, προτύπων και τους ρυθμιστές. Είναι λοιπόν απαραίτητο να υπάρξει μια ενίσχυση της εμπειρογνωμοσύνης που υπάρχει στο δημόσιο τομέα από την Κομισιόν. Κύριε Κλίντς, ειλικρινά. Η ιδέα ενός ταμείου επίλυσης, ενός ταμείου ε, πρόβλεψης κατά κάποιο τρόπο και αντιμετώπιση των κρίσεων. Ξεκινήσαμε να συζητάμε αυτό το θέμα πρόσφατα στη Μαδρίτη, στο ΕΚΟΦΗΝ. με ένα γενικό έγγραφο το οποίο δεν παρουσιάζει αυτό το Ταμείο επίλυση ως μια πανάκια. Είναι μία από τις γραμμές άμυνας, ένα από τα συνολικά εργαλεία που έχουμε, που είναι πολύ περισσότερα, ιδίως στον τομέα της εποπτείας, της εσωτερικής εποπτείας ή εξωτερικής εποπτείας. Θέλουμε να ενισχύσουμε την εποπτεία των διαμεθοριακών πιστοτικών ιδρυμάτων και να δώσουμε και εξουσίες να υπάρξει παρέμβαση πριν από την καταστροφή για να χαλιναγωγηθούν ορισμένες δραστηριότητες, να μην υπάρξει διανομή μερισμάτων σε περίπτωση κρίσης. Και στη συνέχεια όταν μια διαδικασία ε, εποπτείας βλέπει ότι αυξάνονται οι κίνδυνοι, να επιτραπεί η αναδιάθρωση ενός πιστοτικού φορέα προτού καταρρεύσει. Γι' αυτό λέω ότι πρέπει να γίνονται αυτά τα πράγματα χωρίς να πληρώνει πάντα ο φορολογούμενος. Δεν ξέρω λοιπόν κύριε Κλίνης ποιο θα είναι το ύψος αυτού του Ταμείου Επίλυσης και πώς θα λειτουργήσει. Έχουμε ξεκινήσει τη συζήτηση, θα υπάρξει συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων σε αυτή τη συζήτηση και φυσικά δεν μπορώ να ξέρω πόσα χρήματα θα συν, συνενωθούν για κάτι τέτοιο. Ο κ. Γκουλάρ και ο κύριος Γκοζές ξέρουν ήδη πόσο δύσκολα είναι αυτά τα θέματα. Δεν μπορώ να προκαταλάβω λοιπόν πόσα χρήματα θα χρησιμοποιηθούν και πώς θα συλλεγούν. Αλλά δεν μπορεί ο, ο φορολογούμενος να είναι πάντα ο πρώτος που πληρώνει την ύφη. Πρέπει λοιπόν να δημιουργηθεί ένα τέτοιο ταμείο επίλυση σε κάθε μία από τι χώρε μα. Κυρία Σουίνμπερν, ναι. Πρέπει να φροντίσω να είναι συντονισμένα τα μέτρα που παίρνουμε σε ό,τι αφορούν στον αντίκτυπό του. Προσέχουμε πάρα πολύ τι μικρομεσαίε επιχειρήσει και τι συνέπειε για τι μικρομεσαίε επιχειρήσει των ε, ενεργειών μα. Αυτό αφορά και τα παράγωγα, όπου πρέπει να προστατεύσουμε τον τομέα τον βιομηχανικό από τις κρίσεις τις χρηματοπιστωτικές, νομίζω ότι η πρόληψη των κρίσεων θα πρέπει να συντρέχουν με μια βελτίωση της ευκυβερνησίας της επιχειρήσης και όλο αυτό το πακέτο που είναι τμήμα της εργαλειοθήκης πρόληψης των κρίσεων θα πρέπει να λειτουργήσει συντονισμένα και πρόληψη των κρίσεων και καλύτερη ευκυβερνησία και μεγαλύτερη υπευθυνοποίηση των στελεχών και των ηγετών των επιχειρήσεων. Κύριε Μακ, στην οδηγία MIFID. Αντιμετωπίσουμε το θέμα των σκοτεινών δεξαμενών. Δεν έχω να πω τίποτα για την έγκριτη Goldman Sachs. Υπάρχει μια έρευνα που γίνεται από την Αμερικανική δικαιοσύνη, αλλά αν τα γεγονότα αυτά, τα οποία είναι αντικείμενα αυτή τη ανακριτική έρευνα, είναι σωστά, είναι ένα σκάνδαλο αυτό που έγινε. Σκάνδαλο. Έλλειψη ηθικού αναστήματος, έλλειψης ηθικής δράσης με αυτή την τράπεζα η οποία παρέχει χρηματοοικονομικά προϊόντα τόσο πολύπλοκα που δεν μπορεί η ίδια να ελέγξει τη χρήση τους. Αυτό με ενισχύει στη θέλησή μου να ρηφθεί άπλετον φως σε χώρους όπου δεν υπάρχει πάντα φως και που πρέπει να υποχρεθούν να εργάζονται με το μεγαλύτερο επίπεδο διαφάνειας και ελέγχου. Κυρία Μακάρτη, ξέρω ότι υπάρχει κάποια χρονική απόσταση σε σχέση με τους Αμερικανούς σε ό,τι αφορά την εφαρμογή της CRD3. Εγώ θα σας πληροφορήσω επίσης για τα αποτελέσματα της επίσκεψής μου στις ΗΠΑ για το συγκεκριμένο αυτό θέμα, αλλά και επίσης και για τα θέματα καθυστέρησης. Αν υπάρχουν καθυστέρησεις θα πρέπει να εφαρμοστούν οι κανόνες. Κύριε Αποδηματά, αναφερθήκατε στην κατάσταση της Ελλάδος και το ρόλο των φόρων πιστοληπτικής αξιολόγησης που αναφέρθηκα σε αυτόν προηγουμένως. Και εδώ θα πρέπει να εξασφαλιστεί η διαφάνεια για τη μεθοδολογία με την οποία εργάζονται οι φορείς αυτή πιστοληπτικής αξιολόγησης. Και η κυρία Ποδηματά, σας είπα ποια είναι τα συμπεράσματα τα οποία έχω αντλήσει από όλα αυτά που έγιναν. Ήταν μια απόφαση που εγώ σας είχα ανακοινώσει στις 13 Ιανουαρίου πρωτού ξεσπάσει η ελληνική κρίση για τη ρύθμιση του συνόλου των παραγόγων προϊόντων, μεταξύ των οποίων και τα CDS. Και μπορώ να σας επιβεβαιώσω ότι για τα CDS θα αντιμετωπίσουμε το θέμα αυτό συνολικά στο κείμενο για τα παράγωγα προϊόντα του μηνός του Ιουνίου ή Ιουλίου. Και το λέω αυτό τώρα στον κύριο Μπούλμαν που έθεσε ένα ερώτημα σχετικό. Θα δούμε στο ειδικό κείμενο που θα θέσουμε που θα σας δώσουμε τον ε, Οκτώβριο για τον ειδικό ρόλο των CDS όταν αφορούν το κρατικό χρέος, τα κρατικά ομόλογα. Αναφέρθηκε από διάφορους ομιλητές και από την κυρία Φόρ το θέμα των τοξικών στοιχείων ενεργητικού και από την κυρία Οκόνη. Το θέμα αυτό αφορά, ε, αντιμετωπίζεται στο κείμενο για την τίτλοποίηση. Υπάρχει εκεί η υποχρέωση για τις τράπεζες να διατηρήσουν ένα τμήμα των ε, αξιογράφων που εκδίδουν. Κυρία Οκονή, όπως και ο κύριος ε, Μπουλμάν θέσατε το θέμα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και εμείς σε ό,τι αφορά τον αντίκτυπο των μέτρων δίνουμε πάντα μια ιδιαίτερη σημασία στις συνέπειες που θα προκύψουν για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και κύριε Μπούλμαν, μας ενδιαφέρει και η χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που έχουν πρόσβαση στα χρηματιστήρια. Ίσως θα μπορούσαμε να έχουμε ένα χρηματιστήριο που να είναι μια διαδικτύωση τοπικών χρηματιστήριων που να δίνουν μεγαλύτερη πρόσβαση σε χρηματοδότηση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Κύριε Χερκμακ, αναφερθήκατε και εσείς στον αντίκτυπο αυτών των μέτρων. Εμείς έχουμε την ανάγκη να καταμετρήσουμε, αλλά συγχρόνως και να δράσουμε και εκ των υστέρων να αντλήσουμε συμπεράσματα. Στον τομέα αυτό της τραπεζικής ρύθμισης και για τις ε, ασφαλιστικές εταιρείε πρέπει να τα να ακολουθήσουμε αυτές τις κατευθύνσεις για την κυρία Φόρτ. Χρειάζεται ε, περισσότερη υποπτία και σίγουρα κάποιες μορφές συναλλαγών είναι πιο επικίνδυνες από τις άλλες και επομένως θα χρειαστεί καλύτερη υποπτία στο σύνολο του χρηματοπιστωτικού τομέα. Για τον κύριο Ντομένιτσι νομίζω ότι απάντησα για τις γυμνές πωλήσει τον Οκτώβριο θα εκδώσουμε κάποιο νομοθέτημα για τα θέματα αυτά. Αναφέρθηκε επίσης από άλλους ομιλητές το θέμα των ε, φορέων πιστοληπτικής αξιολόγησης και το είπα εγώ σαφώς την προηγούμενη Πέμπτη η Παρασκευή ότι έχουμε ξεκινήσει αυτή την εργασία για τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού φορέα για να αντιμετωπίσουμε ακριβώς το θέμα της ανάλυσης και της εκτίμησης των κινδύνων στα κρατικά αξιόγραφα. Νομίζω θα δώσει προσθέμενη αξία μια τέτοια υπηρεσία και θα δώσει μεγαλύτερη πολυμορφία και ποικιλία στους φορείς, στους φορείς πιστοληπτικής αξιολόγησης. Κύριε Μπουλμάν, θέλετε μεγαλύτερο έλεγχο για τα CDS, θέλετε να είναι υποχρεωτική η εγγραφή των συναλλαγών στα CDS σε μητρώες συναλλαγών, ιδίως όταν πρόκειται για δημόσιο χρέος. Θα κοιτάξω πολύ προσεκτικά τις προτάσεις αυτές, κύριε Μπούλμαν. Και σε σχέση με τις ιδέες του κυρίου Καράς που αναφέρεται προηγουμένως, ο κύριος Κενκέν αναφέρθηκε και στο θέμα των φορέων των μητρών καταγραφής των συναλλαγών αφενός και των φορέων κεντρικού συμψηφίσμου. Αυτό είναι ένα πολύ δύσκολο θέμα, το θέμα της διαλειτουργικότητας των κεντρικών φορέων συμψηφισμού και πολύ τεχνικό. Θα πρέπει να εξετάσουμε πώς μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα να μιλάω για το ρόλο της Ευρώπης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ό,τι αφορά τη δημιουργία φορέων συμψηφισμού. Υπάρχουν σε άλλα μέρη του κόσμου και το ίδιο ισχύει και για τους φορείς συμψηφισμού και για τα μητρώα συναλλαγών, τα trade repositories. Είναι θέμα κυριαρχίας της Ευρώπης και αυτό είναι τμήμα του διαλόγου που έχουμε με τις ΗΠΑ. Θα μελετήσω λοιπόν το θέμα αυτή, το της διαλειτουργικότητας σε τεχνικό επίπεδο, με στόχο, με δύο στόχους, αφενός να έχουμε μεγαλύτερη ασφάλεια και τη σταθερότητα του συστήματος και παράλληλα να μπορέσουμε να διατηρήσουμε ένα επαρκή βαθμό ανταγωνισμού. Για την τοποθεσία στην οποία πρέπει να βρίσκονται αυτοί οι φορείς συμψηφισμού, για μένα είναι σημαντικό η Ευρώπη να έχει τα απαραίτητα μέσα για να συμψηφίσει όλα τα παράγωγα τα οποία βρίσκονται στην αγορά της με έναν τρόπο ο οποίος θα υπόκειται σε εποπτεία και επομένως να έχει και τη δυνατότητα να, να συνδιαλέγεται με τις ΗΠΑ. Δεν έχω λοιπόν κανένα πρόβλημα για το να υπάρξουν τα απαραίτητα ε, μέσα για να έχουμε τους φορείς αυτούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να μπορούμε να συζητούμε με ισορροπημένο τρόπο με τους Αμερικανούς. Πρέπει να έχουν καλή εποπτεία αυτοί οι φορείς και φυσικά να έχουν και επαρκή κεφάλαιο. Θα προχωρήσουμε βέβαια σε μια δημόσια διαβούλευση για τα θέματα αυτά, όπως και πριν από οποιαδήποτε άλλη πρωτοβουλία. Για μένα όμως είναι ένα κεντρικό θέμα αυτό γιατί 80% των συναλλαγών για τα παράγωγα εκφεύγουν κάθε ελέγχου και εποπτείας, κάθε καταγραφής, κάθε συμψηφισμού. Και σας λέω ότι ο στόχος μας είναι να το ανατρέψουμε αυτό και να γίνεται το αντίθετο. Όλα, τα 80% τουλάχιστον να καταγράφονται και να συμψηφίσονται. Γιατί η ευθύνη μας είναι ακριβώς να έχουμε γνώση των πραγμάτων και έλεγχο και πρέπει να έχουμε τα μέσα για να κάνουμε αυτό τον έλεγχο. Σας ευχαριστώ πολύ για την υπομονή σας και την προσοχή σας. Thank you, Commissioner. I'm, I'm sure when you're hearing you thought that that was the maximum pressure you'd have, but I... I... Σίγουρα στην ακρόασή σας θα διαπιστώσετε και τώρα ότι και εδώ υπάρχουν ένα σωρό ερωτήσει και εκεί θα ακούσετε και εδώ δείχνει, αυτό δείχνει πόσο Πολύ δουλειά μένει ακόμα να γίνει. Σας ευχαριστούμε που ήρθατε και σας περιμένουμε τα άλλη φορά.